Mes chers collègues, bonjour. Comme vous pouvez remarquer, je suis en forme. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Γνωρίζετε, είχα κάποιες μικρές περιπέτειες στο Στρασβούργο, αλλά τώρα όλα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι όρθια και θα συνεχίσω να είμαι καλά ε, μέχρι το τέλος της θητείας. Τι έγινε μεταξύ. Κάναμε μια ε, επίσκεψη αποστολή στην Πολωνία. Μας έφερε και μπισκότα ο κύριος Βαντερκόλ. Βαντεκόμπ, Και ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μην καθυστερούμε. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ενακοινώσεις της Προέδρου δεν έχω. Είστε τυχεροί. Ας περάσουμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Να ελέγξουμε την απαρτία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε την α, απαρτία μας και επίσης θα Σα αναφέρω ότι δύο συνάδελφοι, επειδή έχουν ξεχάσει τι κάρτε του, τα ψηφίζουν με διανάτεση τη χειρό. Τρει και ο κύριο Σαλίνη, καλησπέρα. καλησπέρα. Το ECR υπάρχει ένας περισσότερος, ένας παραπάνω. για το ECR βρείτε ποιος δεν θα ψηφίζει. Υπάρχει ένας, μια ψήφος παραπάνω. Γιατί. Α, εσείς ήσασταν. Εντάξει. c'est correct. Ωραία. Είναι όλα σωστά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ξεκινώντας από την έκθεση του κύριου Έρτουκ. Για τις υποδομές που θα πρέπει να δημιουργηθούν για την χρήση εναλλακτικών ε, καυσίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, κύριος Ζήλερ. Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση από την πλευρά του ECR. Είμαστε έξι στην Τραν. Έξι μέλη. Βλέπετε, είμαστε στην σειρά εδώ όλοι καθισμένοι και ο Τόμας στο πάνελ. Τέσσερα τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά. Έξι στο σύνολο. Κύριε Τσίλερ, πράγματι, έχετε έξι μέλη στην Επιτροπή μα, Αλλά εντωμεταξύ δεν έχει αλλάξει το ηλεκτρονικό μα σύστημα, το λογισμικό. Και μου έλεγε ότι υπήρχε ένα υπεράριθμος σε σχέση με τη δύναμη της, των ομάδων. Τώρα και αν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να έρθετε να δείτε την οθόνη του υπολογιστή μου. ερώτηση του κυρίου Τσίλερ, τι εμπιστεύεστε περισσότερο, το λογισμικό ή τη δημοκρατία. Απάντηση της Προέδρου. Πιστεύω στη δημοκρατία, κύριε Τσίλερ. Αλλά τώρα πώς να κάνω την ψηφοφορία. Εάν έχει αλλάξει το μεταξύ ο ρυθμός των μελών και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υπεράριθμη η ψήφος, θα την μετρήσουμε. Θα την προσμετρήσουμε. Είδατε, σας έπεισα ότι πιστεύω με τη δημοκρατία και όχι τα ρομπότ. Έχει εγκριθεί και η συμβαστική 3. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Ε, όχι, ζητείτε να ελέγξουμε για την 35. Ψηφίστε παρακαλώ. 53. Ε, πέρας ψηφοφορίας ανακοινώνει η πρόεδρος. Έχετε δίκιο, κύριε Σαλίνη. Εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ. Συμβαστική 3. Κατά. Αποχές. Α, δεν ήταν ξεκάθαρο. Ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για τη συμβαστική 3. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται η συμβιβαστική 3. Κυρία Μπιλμπάο, τι ψηφίσατε, υπέρ ή κατά. Υπέρ. Άρα 17 υπέρ. Και ε, ε, ε, εσεί μεταξύ βρήκατε την κάρτα σα, επομένω η συμβιβαστική τρία εγκρίνεται αν συμπεριλάβουμε και την ψήφο τη κυρία Μπιλμπάου. Είπατε κύριε Αρτούγκα. Και μέτρησα και τις έξι ψήφους του ECR, να το πω και αυτό. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV35 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Τι κάνει το ΕΛΚ. Για ξυπνήστε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Τροπολογία 85, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές Δεν είναι ξεκάθαρο. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 68. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ξεκάθαρα. Να σηκώνετε ψηλά το χέρι, παρακαλώ, για να μην χρειάζεται αυτό. Ωραία. Πάμε κατευθείαν στην NV19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται μάλλον. Ναι, ναι, εγκρίνεται λέει η πρόεδρος. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τοπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 15 υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Α ελέγξουμε. Για την τροπολογία 3 ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρα ψηφορία, εγκρίνεται. Και η κυρία Μπιλπάου σημειώνω, είναι υπέρ. 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ήτρε. Α. Υπέρ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 Συμβιβαστική 17. Ευχαριστώ κύριε Νταλόν που με... Το θυμήσατε. Υπέρ για 17. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 15. υπέρ ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 25. 25. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές το ΕΛΚ τι ψηφίζει υπέρ είστε ψηφίζετε υπέρ α ωραία να ξαναψηφίσουμε λοιπόν 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Allez, je ferme le vote. ψηφοφορίας και η κυρία Μπιλπάου ψηφίζει υπέρ. Άρα 29 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, 6 εποχές. Συγχαρητήρια κύριε Ερτούκ, εγκρίνεται η εκθεσή σας. Allez, nous avec Συνεχίζουμε την πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη περίγραφος 2021 ε, με 2027. Πρόκειται για γνωμοτότηση προς την Επιτροπή Ήτρα και ο εισηγητής μας και η κυρία Κλούνα. Καλημέρα σας. Αν παρακαλώ θέλετε να κάνετε συζητήσεις έξω από την αίθουσα. Έχει το λόγο η κυρία Κλούν. Μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027 πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής προς την Επιτροπή Βιομηχανίας. Καταρχάς, καλώς ορίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίσει αυτό το πρόγραμμα με βασικό στόχο να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και ευρωπαϊκής κοινωνίας. Πολύ ευπρόσδεκτο και θα πρέπει να φροντίσουμε να προωθήσουμε την τεχνική επανάσταση προκειμένου η οικονομία μας να είναι επαρκώς προετοιμασμένη για τις νέες αυτές προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Να προωθήσουμε μια βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη. Αυτό έχει και ως σκοπό το πρόγραμμα αυτό. Είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό ψηφιακό πρόγραμμα και θα ενώσει όλες τις περιοχές της Ένωσης. Από πλευράς ε, μεταφορών, νομίζω ότι το βασικό στοιχείο της κυβερνοασφάλειας είναι ευπρόσδεκτο εδώ στην έκθεση και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα ασφάλεια στον τομέα μεταφορών, μιας και όλα αυτά θα είναι όλο και πιο πολύ διασυνδεδεμένα και το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς οι μεταφορές θα καταστούν όλο και πιο διασυνδεδεμένες. Υποστηρίζω λοιπόν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου σε ψηφιακό επίπεδο να υπάρχει επιτέλους ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να θίξω σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά και τα αυτοκινούμενα οχήματα τα οποία όλο και πιο πολύ προωθούνται. Θα πρέπει να διευκρινίσει, θεωρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανόνες ασφάλειας και ευθύνη σε ό,τι αφορά τη θέση σε εμπορία. Και επίση ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι κατάλληλο και για νεοφύης και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να καταλάβουν ένα καλό μερίδιο της αγοράς. Το πρόγραμμα επίσης θα πρέπει να λάβει υπόθεση, υπόψη και το δυναμικό της ψηφιοποίησης σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους, τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και τέλος, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξασφαλίσει μία συνεργεία και με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης όπως το ΣΕΦ2 για παράδειγμα για να υπάρξει καλύτερη δυνατή υποστήριξη προγραμμάτων και έργων που έχουν διασυνοριακό διατομιακό χαρακτήρα και να υπάρχει καλή χρήση α, πόρων για προς των πολιτών. Προσβλέπω λοιπόν να ακούσω και τους άλλους εισηγητές και να κατακτήσουμε τελικά μια κοινή τοποθέτηση Επιτροπής Μεταφορών και Βιομηχανίας. Ελπίζω να είναι επικοδομητικές οι συζητήσεις, όσο επικοδομητικές ήταν και για την προετοιμασία της χρωματοδότησης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κλούν, λέει η Πρόεδρος, οι σοσιαλιστές τώρα. Ο κύριος Καπούτο δεν είναι παρόν. Ποιος θα πάρει το λόγο εξ ονόματός του. Κανείς. Καλά. Ο κύριος Τοντανόφσκι. Έχει το λόγο. Α, ο κύριος Νουτόσκι. Κοιτάξτε, είναι στη θέση του κύριου Τουζανόφσκι, παίρνει το λόγο. Ο σκιώδης μας εισηγητής, ο κύριος Τουζανόφσκι, έφυγε, πήγε στην Επιτροπή Ήτρε, που είναι η κύρια επιτροπή του και μου ζήτησε να παρουσιάσω το μήνυμα το οποίο έχει να μεταφέρει. Καλώς ορίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς και αναγνωρίζει ότι είναι έξοχη η βάση του κειμένου της εισηγητρίας για την περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου. Θεωρεί όλα αυτά ότι θα μπορεί, υπάρχει κάποια περιθώριο βελτίωση σε κάποια σημεία. Καταρχάς, το θέμα της κυβερνοασφάλειας παίζει φυσικά βασικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να προωθηθούν και άλλες, ε, άλλες στόχοι, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Κατά δεύτερον, ο εισηγητής τονίζει σωστά την ανάγκη να υπάρξουν συνέργειες και με άλλα προγράμματα και με άλλα ταμεία. Τονίζει επίσης και το νέο πρόγραμμα και το διάστημα που καλύπτει τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο και άλλα επιτυχή προγράμματα. Και τέλος, ε, ο σκιώδης μας πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές, ε, τους ψηφιακούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και με τις χώρες. Θα καταθέσει ενδεχομένω σχετικέ τροπολογίες και προσβλέπει σε μια επικοδομητική συνεργασία με την κυρία εισηγήτρια και τους άλλους σκιώδες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ντίρντε Κλούν για την δουλειά της, τον θαυμάσια δουλειά. Περιμέναμε αυτή την έκθεση εδώ και δέκα χρόνια. Μία τέτοια πρόταση, αν υπήρχε ο πλευρά Κομισιόν πριν από 10 χρόνια, νομίζω ότι ο ψυχιακός κλάδο στην Ευρώπη θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τώρα. Αλλά τέλο πάντων, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ε, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και τις τροπολογίες α, της εισηγήτριας. Ε, οι πέντε ειδικοί στόχοι αντιστοιχούν στους βασικούς άξονες ε, παρέμβασης της Κομισιόν. Επομένως, βρίσκουμε και τις παρεμβάσεις στον τομέα των μεταφορών, καθώς και στα επιπρόσθετα και καινοτόμα θέματα ε, των αυτόνομων οχημάτων και της μεταφοράς μέσω σιδηροδρόμων. Υποστηρίζουμε πολύ καλά την ένταξη των αυτόνομων οχημάτων στις δράσεις που υποστηρίζει το πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τις συνέργειες ε, μεταξύ μεταφορών και τηλεπικοινωνιών ε, και ειδικά στα δίκτυα. Επομένως, η διάρθρωση, όπως υπόθηκε με άλλα προγράμματα, η σύνδεση με άλλα προγράμματα, ε, μας απασχολούν και γι' αυτό θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες, όχι πολλές, λίγες, γιατί έχω ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με την πρόταση της Κομισιόν. η οποία δεν έχει πολλέ αντιδράσει ούτω ή άλλω από βουλευρά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Thank you, Chair. Εκπροσωπώ την Jill Evans, η οποία μου ζήτησε να σας πω ότι καλωσορίζει το σχέδιο γνωμοδότης της εισηγήτριας και θέλει να το ενισχύσει περαιτέρω με τα εξή σημεία προστασία δεδομένων και ιδιωτική σφαίρα, διατήρηση και δημιουργία ε, θέσεων ε, απασχόληση υψηλή ποιότητα, υποστήριξη των ΜΜΕ και αύξηση τη ψηφιοποίηση με εστίαση στην διαχείριση τη ε, κινητικότητα και πράσινη επιμελητία, ούτω ώστε να υποστηρίξουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών. Είστε πολύ αποτελεσματικό. Μπράβο σα. Και στραφούμε προ την Κομισιόν και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μιέλοφ. Μιχάηλοφ. Η Κομισιόν, εν πάση περιπτώσει, έχει το λόγο. Ούτως ή άλλως είχαμε προτείνει τα, το όραμά μας, αλλά καλύτερα να τα πω αγγλικά γιατί γαλλικά ε, δύσκολο. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που ακούστηκε, είναι ένας ειδικό στόχος Έχουμε διάφορους τομείς που θα θέλαμε να εφαρμόσουμε, να χρησιμοποιήσουμε την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης υπάρχει ένας στόχος για τις έξυπνες πόλεις ε, και θα εστιάσουμε στις μεταφορές και στην ενέργεια στα πλαίσια των έξυπνων πόλεων και θα θέλαμε και να απεικονίζονται αυτές, ε, αυτοί οι άξονες, αλλά να υπάρχουν και συνέργειες ανάμεσα αυτούς τους δύο άξονες. Γιατί έχουμε εφαρμογές οι οποίες αφορούν και τους δύο. Οποιοδήποτε ε, σύστημα, αυτόνομο σύστημα μεταφορών μέσα στην πόλη θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια αστική πλατφόρμα. Γι' αυτό στο στόχο αυτό έχουμε προβλέψει την ε, μαζική ανάπτυξη ε, τέτοιων πλατφορμών για τις πόλεις, για τις έξυπνες πόλεις που θα διαχειρίζονται διάφορα συστήματα που αφορούν τις πόλεις είναι οι πιο κοσμοβρυθείς ε, περιοχές ε, οι πόλεις, όπου ε, έχουμε τον μεγαλύτερο πληθυσμό, ΑΕΠ και τα λοιπά, αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά και τις προαστιακές περιοχές. Ε, σας παραπέμπω ειδικά στα αυτόνομα οχήματα, ειδικά σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα των προαστιακών περιοχών. Μία μικρή ερώτηση προς την Κομισιόν, λέει η Πρόεδρος. Εάν θέλουμε να υπάρχει παντού σύνδεση, παντού ψηφιοποίηση, ε, τι κάνετε για το 5G, για τις υποδομές. Ε, θα αναπτύξετε σε όλες τις υποδομές το 5G. Να απαντήσω. Το, οι υποδομές 5G, ε, ε, αυτά τα δίκτυα αφορούν το SAFE. Είναι το πρόγραμμα SAFE. Εδώ μιλάμε περισσότερο για τους ε, διαδρόμους, τις μεταφορές και την ανάπτυξη διαδρόμων ε, που θα χρησιμοποιούν το 5G. Το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη δεν αφορά τα δίκτυα και την ε, ευρυζωνικότητα και το 5G, αλλά τις τρεις βασικές τεχνολογίες που έχουμε εντοπίσει, που είναι σημαντικές για το μέλλον, το ψηφιακό της Ευρώπης. Νοασφάλεια, και AI, τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν ε, στις μεταφορές, κυρίως τα αυτόνομα οχήματα, οι ευκαιρίες που προέρχονται από τεχνητή νοημοσύνη και από την κυβερνοασφάλεια. Σε αυτούς τους τομείς εστιάζει το πρόγραμμα, όχι στο 5G. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση. Γιατί πραγματικά, κυρία Κλούνα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έκθεσή σας. Μιλάτε για τεχνητή νοημοσύνη. Μπορείτε να μου δώσετε έναν ορισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να καταλήξει σε έναν ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να σας δώσω έναν ορισμό, αλλά όχι τώρα, θα το αποφύγω. Γιατί θα ήταν τελείως προσωπικός ορισμός και δεν θα ήταν σωστό σε αυτή τη φάση. Έχουμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για την τεχνητή νοημοσύνη που άρχισε τι συνεδριάσει. Έχει Έχει συνεδριάσει μόνο μια φορά μέχρι στιγμή, αλλά θα καταλήξει μια έκθεση για διάφορα θέματα και το πρώτο ερώτημα που θα τους απασχολήσει και ήδη τους απασχολεί είναι ακριβώς ο ορισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Θα καταλήξουμε σε ένα σαφέστατο ορισμό σε λίγους μήνες. Υποτίθεται ότι η ομάδα αυτή θα ολοκληρώσει αυτό το θέμα στο τέλ, στα τέλη της χρονιάς. Και εγώ ήθελα αυτό, να, αυτό το πράγμα, να έχω δηλαδή έναν ορισμό μέχρι το τέλος του 18. Η εισηγήτρια για να κλείσει την έκθεσή της. Ευχαριστώ και τους κοιόδης συγητές. Έχουμε πολλές, πολλά θετικά στοιχεία, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Σας ευχαριστώ και σας Πρόεδρε για τις ερωτήσεις σας που μπαίνετε σε αυτά τα θέματα. Είμαι έτοιμη να συζητήσω με βάση τις προτάσεις και τις τροπολογίες που θα κατατεθούν στον επόμενο γύρο. Θα συζητήσω και με τους κοιόδης εισηγητές και είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό για την Επιτροπή μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε εισηγήτρια για, τις, ε, για σας. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 5η 27 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Να συνεχίσουμε. Να σας ζητήσω το εξής. Ο κύριος ε, ο Βάντε Κάμπ θέλει να συνεχίσει τώρα ή να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να συνεχίσουμε. Μάλιστα. Έχουμε πρόταση κανονισμού ε, για το πρόγραμμα InvestEU. Είσαστε εισηγητής, κύριε Βαντεκάμπ. Έχετε το λόγο. μικρόφωνο, κύριε Βαντεκάμπ. Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι άλλο θέλω να αναφέρω. Θέλετε να σας μιλήσω για την αντιπροσωπεία στην Πολωνία ή θέλετε να το κάνουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Τι θέλετε. Θα το συζητήσουμε στους συντονιστές άμα θέλετε, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα, ευχαριστώ. Αυτό για να ξέρω που βρίσκομαι. Πρόεδρε, λοιπόν, σήμερα μιλάμε για το νέο πρόγραμμα Invest EU. Invest. Επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το μεταμεταφορών πρόκειται για την συνέχεια του ΕΦΣΙ του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Προγράμματος. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επενδυτικό εργαλείο λοιπόν, όπου η Επιτροπή Ήτρε και Τραν θα έχουν κοινή αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά το άρθρο 54 οι καθήλυνα αρμόδιες είναι η Επιτροπή Προπολογισμών και Ελέγχου του Προπολογισμού, αλλά σε 3, 4 και 7 και στα προσαρτήματα, σε 1, 2 και 3, έχουμε α, ε, κοινή αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 54, όπως σας είπα. Πρόεδρε, υπήρχε επί μακρόν μία αμφιβολία για την επιτυχία του ΕΦΣΥ σε ό,τι αφορά τον τομέα των μεταφορών τουλάχιστον. και έχουμε 24 δισεκατομμύρια φτάσει σε ό,τι αφορά τι επενδύσει μέχρι την άνοιξη του 2018. Και αυτό συνοδεύεται και με την επένδυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο πολλαπλωσιαστικός λοιπόν παράγοντας είναι τριπλάσιο ουσιαστικά σε σχέση με το αρχικά επενδυμένο ποσό. Τώρα περνάμε λοιπόν στο InvestEU. Είναι σαφές αυτό για όλους σας ότι όλα αυτά συγκαταλέγονται στις γενικότερες διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο οι οποίες γίνονται σε υψηλό βαθμό επίπεδο. Έχουμε και την προσέγγιση μέσω του Συνδέατα στην Ευρώπη, το ΣΕΦ, αλλά έχουμε και το InvestEU πλέον λοιπόν. Και εδώ θα έχουμε μία εγγύηση 38 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο θα οδηγήσει σε επένδυση 15,2 δις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τα επαναλάβω. Επένδυση 15,2 δις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εγγυημένη επένδυση σε ύψος 38 δισεκατομμυρίων Στο Investing in You λοιπόν, κοιτάμε κυρίως τις βιώσιμες υποδομές. Αυτή η προσέγγιση μας απασχολεί. Sustainable Infrastructure Window στα αγγλικά. Εδώ έχουμε 11,5 δις ευρώ. Πρόκειται για ποσά τα οποία μπορούν να έχουν μεγάλο αντικτύπο λοιπόν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να αντιληφθούμε λοιπόν ότι το InvestEU είναι μία απλοποίηση των κανόνων TNT γιατί ε, πρόκειται για ομαδοποίηση των οικονομικών κονδυλίων τα οποία συναπαρτίζουν το ΣΕΦ μέχρι τώρα. Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στην πολιτική για το κλίμα και αυτό προφανώς δεν προκαλεί έκπληξη γιατί όλοι παρακολουθήσαμε την COP21 αλλά παράλληλα δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση και στην ασφάλεια και στις ευκαιρίες απασχόλησης σε ό,τι αφορά τους απασχολούμενους στον τομέα των μεταφορών αλλά και στον τουρισμό. Πρόεδρε, τώρα ε, σημαντικά είναι και τα προσαρτήματα Ξέρετε ότι συχνά έχουμε στο κείμενο το διδακτικό τους ε, βασικούς κανόνες, αλλά οι πικάντικες λεπτομέρειες κρίνονται στα παρατήματα. Και είναι σημαντικό λοιπόν να τις προσέξουμε. Για παράδειγμα, πιο πολύ προσοχή για τα αυτοκινούμενα, αυτοκινούμενες λύσεις. Επίσης, μεγαλύτερη σημασία για τα έργα τα διασυνοριακά cross-border. Παράλληλα να δείξουμε προσοχή για να υπάρξει γεωγραφική ισορροπία μεταξύ κρατών μελών. Επίσης, μεγαλύτερη προσοχή στο τουρισμό, γιατί ο τουρισμός ε, πλέον ε, αποτελεί μεγάλο οικονομικό κλάδο. Παράλληλα, πιστεύω ότι το InvestEU θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση μεταξύ των μεταφορών και της ποιήψης. Το ότι οι επενδυτικοί στόχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν βιώσιμες υποδομές τουλάχιστον κατά 50% στα πλαίσια της πολιτικής για την προστασία του κλίματος. Έχουμε τρία σημεία στα οποία ασκούμε κριτική. Καταρχάς, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αλλάξει την διαχείριση των προγραμμάτων αυτών σε σχέση και με το ΕΦΣΥ. Στο ΕΦΣΥ μεγάλο ρόλο έπαιζε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα πλέον αυτή την αρμοδιότητα φαίνεται ότι την αναλαμβάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ φοβάμαι, φοβάμαι Προέδρα, γιατί θεωρώ ότι θα προκύψει ένα διπλό σύστημα γραφειοκρατίας. Γραφειοκρατία και της ΕΤΕΠ και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα θέλω να μας το εξηγήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το έχει φανταστεί. Ύστερα, να προσέξουμε, γιατί στο InvestEU σημαντικό ρόλο παίζει η ανανέωση και προστιθέμενη αξία. και όχι ο διπλασιασμός τέτοιων ε, προγραμμάτων. Θέλουμε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ ενεργείας και ψηφιακής διάστασης προφανώς. Και θεωρώ την επόμενη Τετάρτη, την Παραπέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου, ε, θεωρώ ότι θα γίνει η πρώτη παρουσίαση και η παρουσίαση των τροπολογιών για αυτό το πολύ ενδιαφέρον στο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Winfrom και να ξεκινήσει λοιπόν πάρα αυτά η συζήτηση. Το λόγο έχει... Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή του κειμένου και τον κύριο Φοντεκάμπ για την έκθεση. Και όντω το μέσο των μεταφορών αποτελεί το τομέα κλειδί για να πετύχουμε τις δεσμεύσεις μας ε, τη συνθήκη του Παρισιού, τους κλιματικούς μας στόχους. Και επίσης σημαντικό είναι να υπάρχουν ε, αντίστοιχε ε, δημόσια κίνητρα. Εδώ όμως θέλω να το μείνω ότι θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη εκπροσώπηση για το τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει να προσέξουμε ο τομέας της κινητικότητας και η αλλαγή της κινητικότητας να μην φορτωθεί στις πλάτες του φορολογούμενου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου αυτές οι λύσεις να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε οικονομικά αδύναμες κοινότητες. Το κόστο λοιπόν τη κινητικότητα αυτές δεν θα πρέπει να βαρύνει του πολιτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία τη, ε, θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει σωστή επένδυση. Ω τώρα η Ευρώπη κινείται προ την λάθος κατεύθυνση όπω είδαμε στο θέμα των διοδίων για τα φορτηγά και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτή η αλλαγή στι μεταφορέ να μην θεωρηθεί μόνο ένας πολιτικός στόχος και ένας στόχος των μεταφορών. Είναι και κοινωνικό θέμα. Άρα δίκαιη άμα, κατανομή των βαρών. Χαίρομαι και προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή. Και εγώ και η ομάδα μου θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ Ο κύριος Λοντόφσκι έχει το λόγο. Bardzo Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τον εισηγητή, για την προετοιμασία του κειμένου. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία αυτού του νέου εργαλείου, το οποίο θα ομαδοποιήσει πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής χρησιμοποιούμε στην Ένωση. Γιατί έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με εναρμόνιση των διαφορετικών διαδικασιών και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε και μια καλύτερη σχέση με τους επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιήσουμε καλύτερα όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο των ε, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και των προγραμμάτων για την περιφερειακή συνοχή. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή για τη σημασία αυτών των θεμάτων. Θα πρέπει το InvestEU να υποστηριχθεί έτσι ώστε να είναι στο ίδιο ύψος με το εύση. Δεν θεωρούμε ότι είναι απλώς μια συνέχεια του Connecting Europe, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το InvestEU για να επενδύσουμε στην ασφάλεια των δρόμων και άλλες τέτοιες σημαντικές προτεραιότητες. Κατά την άποψή μα σε αυτό το τομέα η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να βελτιωθεί. Ένα μεγάλο θέμα για τους επενδυτές είναι ότι το InvestEU καλύπτει το 50% της επένδυσης σε κάποιες υποδομές. και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η σύνδεση αυτή τη πολιτική για την ανανέωση των υποδομών με την πολιτική μα για τη βιώσιμη ανάπτυξη γενικώ. Πιστεύω ότι εάν το ποσοστό πήγαινε από 50% στο 20% θα είχαμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε περισσότερες, περισσότερα έργα και επίσης διευκρίνησε ο κ. Βαντεκάμπ ότι πλέον θα είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό δεν είναι λογικό γιατί η συνεργασία, η λειτουργία ε, αυτών των προγραμμάτων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Επενδύσεων ήταν πολύ ικανοποιητική. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε και την εξειδικευμένη γνώση που έχει συσσωρευτεί σε αυτούς. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Βαντερκάμπ για την προετοιμασία του κειμένου και θα προτείνουμε και από τη δική μας την πλευρά τροπολογίας. Για τους πρασίνους. Όχι, ζητώ συγγνώμη. Κάποιον. Ε, κύριε Ρικέ, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν... Κατάλαβα ότι έπρεπε σε εσάς να δώσω το λόγο. Κύριε Ρικέ. Βιμ, κύριε Φαντερκάμπ, σας ευχαριστώ για αυτό το πολύ καλό προσχέδιο της νομοδότησης. Υποστηρίζω τις προτάσεις σας. ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στη βελτίωση του μηχανισμού, την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί στον τουρισμό, κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε στο στοιχείο σε αυτές τις αυτά τα εργαλεία. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη συζήτηση για τις μειώσεις που γίνονται σε κάποιες προτεραιότητες όπως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και το, η, και η, συντήρηση και το upgrading των υποδομών είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις οδικές μεταφορές, για να καταπολεμήσουμε την ατμοσφαιρική ρήπανση από τις οδικές μεταφορές. Επίσης ήταν χρήσιμο αυτό που ακούσαμε σε σχέση με το παράρτημα 2, που είπατε για τις πικάντικες λεπτομέρειες. Δηλαδή, στο παράρτημα 2 βλέπει κανείς ότι θα χρειαστούν παρεμβάσεις ε, για την αξιοποίηση των αλλακτικών καυσίμων, για ε, ε, τα, αεροδρόμια. Μήπως επίσης θα ήθελα καλύτερο να αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα στα αυτόνομα α, οχήματα Επίσης, ίσως έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην μετάφραση στο σημείο στο οποίο αναφέρεστε στη διαφοροποίηση. Πιστεύουμε όμως ότι όποιες παραβάσεις στα δίκτυα θα πρέπει να περιοριστούν σε αυτούς τους τομείς που αναφέρονται στο παράρτημα. Κάτι μεγαλύτερο θα ήταν δύσκολο να γίνει στην πράξη. Τώρα, είναι ουσιαστικό θέμα συζήτησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προέλευση των κονδυλίων, παρόλο που αυτή τη στιγμή συζητούμε για τις μεταφορές και ίσως να μην είναι αυτό το, το θέμα, αλλά είναι σημαντικό. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των προγραμμάτων. Θα ήθελα να χαιρετήσω το γεγονό ότι η διαχείριση των προγραμμάτων πλέον δεν θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Επενδύσεων, αλλά από μια επιτροπή ειδικών επιρρογνωμόνων ε, υπό τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό το χαιρετίζω και δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο Λοτόφσκι, επειδή εμεί δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από το έργο που έκανε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί αυτό. Με όποια διαδικασία και να ακολουθείτε, όποια μάλλον ε, διαδικασία και αν είχε ακολουθηθεί, κατέλεγε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο σημαίνει ότι πολύ συχνά είχαμε μείωση των δημόσιων, ε, της, της, της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένα θέματα. Ήταν έτοιμα λοιπόν να αλλάξει και να βελτιωθεί ο τρόπος διακυβέρνησης και χαίρομαι για αυτή την αλλαγή που έγινε, που διευκρινίζει ε, και ξεχωρίζει μάλλον το, το, τις ε, αρμοδιότητες του καθενός, της διαχείρισης του προγράμματος αφενός και της ε, λήψης της απόφασης αφετέρου. Επίση, χαιρετίζω το γεγονό ότι έχει μεγαλύτερη δημοσιότητα πλέον λάβει το θέμα αυτό και στι πλατφόρμες του Συμβουλίου. Του στόχου βέβαια του προγράμματο θα πρέπει κατά την άποψή μου να του συζητήσουμε περισσότερο και πιο, και πιο διεξοδικά. ο μηχανισμός αυτός ήταν ήδη πολύ σημαντικός, τώρα γίνεται ακόμα καλύτερος, πιο απλουστευμένος καλύτερη διακυβέρνηση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε περισσότερη προστιθέμενη αξία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζω λοιπόν την ε, έκθεση, την προσχέδιο της έκθεσης του κ. Φαντερκάμπ και θα, προσ... θα προστείνουμε και εμείς διάφορες τροπολογίες. Ευχαριστώ και τώρα οικολόγοι. Ε, εγώ ή ο κύριος Κίστελόρ. Εσείς. Sur budget, vous voulez que je le fasse ou vous le faites? γνωμοδότηση του προπολογισμού. Όχι, όχι, έκανα λάθο, λέει ο πρόεδρο, για το InvestEU. Να μιλήσετε εσεί ή εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Βαντενκάπ για την ε, προσπάθειά σας. Η βασική μας ανησυχία είναι ότι οι επενδύσεις και η εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού καθώς και τα δάνεια θα πρέπει να εξασφαλίσουν ε, μια καλύτερη ισορροπία. Καλύτερη δηλαδή ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλη και στις ε, ζημίες. Τι σημαίνει ότι τα κέρδη δεν θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν και οι ζημίες δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά της κοινωνίας. Ειδικά όταν μιλάμε για το δημόσιο κορβανά. Εδώ η τροπολογία σας τρία στο σχέδιο γνωμοδότησης είναι σχετική τροπολογία για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, όταν μιλάμε για επενδύσεις κατά προτεραιότητα, χρειάζονται οπωσδήποτε τέτοιες ε, επενδύσεις και θα πρέπει να συνοδεύονται από πραγματική πρόοδο, δηλαδή έργα. Στους πολύ συγκεκριμένους στόχους τώρα, τους οποίους ε, συζητάμε. Έχουμε στόχους για το κλίμα, κύριε Βαντεγκάμ, το ξέρετε, και θα πρέπει να δούμε αν αυτό το σχέδιο ε, εντάσσεται στους στόχους του Παρισιού και στο στόχο της μείωσης ε, των αερίων του διοξείδου του άνθρακα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να μειώσουμε στο σχέδιο αυτό ε, έκθεση τη σημασία του πώς θα ενσωματώσουμε το εξωτερικό κόστος και θα προλάβουμε τις επιπτώσεις. Κύριε Βάντεν Κάμπ, βάλατε τον τουρισμό σας. Ευχαριστώ γι' αυτό στο σχέδιο γνωμοδότησής σας. Στην αρχή το είχαμε εντελώς αγνοήσει αυτό το θέμα. Θα πρέπει επίσης να καλύψουμε και αυτό το θέμα ε, στα έργα και θα πρέπει να είναι προς όφελος και των τουριστών αλλά και των κατοίκων που υποδέχονται αυτούς τους τουρίστες. Αυτό το, το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως και ένα πράγμα το οποίο δεν κατάλαβα πολύ καλά κύριε Σιγητά και δεν συμφωνώ εδώ με την άποψή σας γιατί λέτε και θα ήθελα κάποιε διευκρινήσει από αυτού, έτσι. Ε, τονίζεται λοιπόν την εξή ιδέα, ότι το λιγότερο από το 5% των επενδύσεων θα πρέπει να συνεισφέρουν στους κλιματικούς στόχους και τους περιβαλλοντικούς στόχους. Δεν συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χικέ ότι θα πρέπει να μας εξηγήσετε το σημείο αυτό. Δεν θέλετε. Ναι ή όχι, θα μου το εξηγήσετε. Δεν, συμφ... Δεν συμφωνείς με τον ε, Ντομινίκ Ρικέ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι. Ο κύριος Ρικέ είναι πολύ οικολόγος. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά εγώ σας το λέω, για να σας φωτίσω. Α, από σήμερα έγινε οικολόγος. Λοιπόν, να μου εξηγήσετε αυτή την επιλογή για να μπορέσω να συζητήσω και τις συμβαστικές ιδέες. Η κυρία Ροβονταλόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης που μας παρουσιάζεται για το πρόγραμμα InvestEU με στόχο να αντικαταστήσουμε το παρόν FC Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει πολύ ενδιαφέρουσες και κατάλληλες προτάσεις για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει ε, προγράμματα μεταφορών. Υποστηρίζω όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για τα παραρτήματα για να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή του προγράμματος στη χρηματοδότηση των συστημάτων RTMS ε για το ε, για τους ιδεοτρόμους, εναλλακτικά καύσαμα για και κυρίως ε, βιώσιμη κινητικότητα. Θα πρέπει το παγκόσμιο προγράμματα, ε, δίκτυο του RTT ε, να συμπεριληφθεί, γιατί δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο ε, τους βασικούς διαδρόμους κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να χρηματοδοτούμε και έργα τα οποία συνεισφέρουν ε, σε μια εδαφική συμμετοχή των πιο απομακρυσμένων περιοχών στα δίκτυα. τώρα, το 50% ε, που θα πάει στους ε, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους δεν είναι επαρκές. Το 50% θα πρέπει να γίνει 60% όπως και στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την ε, διασύνδεση. Τέλος, θα ήθελα να συνεχίσω μια συζήτηση που έγινε όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε τα εύση το θέμα της ε, δημοσιονομικής ευελιξίας. Το πρόγραμμα Investing You δεν θα πρέπει απλώς να επικεντρωθεί στις ε, ιδιωτικές επενδύσει, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετήσει και τη δημόσια επένδυση. Χωρίς δημόσιες επενδύσει, μαζικές δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε τους ε, στόχους μας ό,τι αφορά την οικονομική μετάβαση, οικολογική μετάβαση. Θα προτείνω να βγάλουμε το δημόσιο έλλειμμα, τα δημόσια έλλειμματα ε, από την ε, συγχρηματοδότηση που συνεισφέρουν στην υλοποίηση των κλιματικών και ε, περιβαλλοντικών στόχων στα πλαίσια του InvestEU. Κύριε σας ευχαριστώ για την πρόταση, κύριε Σιγητά. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι να δώσουμε έμφαση στις διασυνοριακές περιοχές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι οι πιο ευπαθείς. Θέλουμε να συνδέσουμε την Ευρώπη και οι διασυνοριακές περιοχές είναι πάντα εκείνες που χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις. Κατά την άποψή μου λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και αυτό, αλλά και το θέμα της γεωγραφικής ισορροπίας λοιπόν. Γιατί στους διάφορους διαγωνισμούς και διάφορες ε, προκηρύξεις υποβολής ε, για την ε, υποβολή αιτήσεων ε, ενδιαφέροντος. Μερικές φορές το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, ο τουρισμός. Κάθε χρόνο ε, αυξάνεται η προσοχή που δίδεται σε αυτό το τομέα που ούτω ή άλλω είναι και θέμα αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα. Κάποιε άλλε παρατηρήσει. Ξέρουμε ότι η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι επενδύσει δεν είναι επαρκή σήμερα για να ανταποκριθούμε στι προκλήσει οι οποίε ε, υπάρχουν και θα υπάρχουν στο μέλλον σε ό,τι αφορά την ανεργία, κοινωνικέ επενδύσει ή κλιματικέ αλλαγέ. Υπάρχει μια δυσκολία πρόσβαση στη χρηματοδότηση ακόμα και σήμερα. Και αυτό εμποδίζει την ενεργοποίηση διαφόρων προγραμμάτων και την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει η Ευρώπη στον εαυτό τη. Ίσως χρειάζονται λιγότεροι κανόνε, αλλά οι κανόνε αυτοί θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Πέρα από ένα πλαίσιο προγραμματισμού πιο ευέλικτο, πρέπει να υπάρχει και σταθερότητα. Το InvestEU νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να δώσουμε μια όθηση στις δημόσιες επενδύσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις, ειδικά στον τομέα των μεταφορών. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει επίσης να υλοποιούν του κλιματικού στόχου, προφανώ. αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την κοινωνική διάσταση. Τέλο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιε είναι ποιοι είναι οι τομεί παρέμβαση του προγράμματο. Δεν θα πρέπει να περιοριστούν στην διατήρηση των ισχύων των, των, των ισχυουσών υποδομών. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Ευχαριστώ και στρέφουμε τώρα προ την Κομισιόν. Έχω την χαρά να έχω μαζί μου εδώ την κυρία, μαζί μας την κυρία Έστερ Γκόγκερ. Ε, καλώς ήρθατε. Και σας δίνω το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε με προσοχή το σχέδιο της έκθεσης του ΙΣΕ, γιατί και άκουσε με προσοχή επίσης τη σημερινή συζήτηση. Υπάρχουν διάφορα σημεία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνοι με τις παρατηρήσεις που έγιναν και υπάρχουν και διάφορα άλλα σημεία. Εν, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ε, τα σχόλια ε, θα πρέπει να μπουν πιο πολύ στα, πιο πολύ στα investment guidelines, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις επενδύσεις που θα ακολουθήσουν σε μετέπειτα χρονική στιγμή και σε άλλα σημεία υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες θα εξετάσουν ε, πιο συγκεκριμένα το θέμα των κλιματικών στόχων. Στα θέματα διακυβέρνησης, οι αλλαγές σε σχέση με το ΕΦΣΥ δικαιολογούνται από δύο αιτίες. Καταρχάς, ανοίγει το θέμα της εγγύησης, υπάρχει πρόσβαση στην εγγύηση. Η ΕΤΕΠ θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό εταιρό συνεργασίας, αλλά αναμένουμε και άλλους ε, ε, εταίρους όπως ε, η BID. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αποτυπώνεται σε μια πιο ανεκτική πρόσβαση και κατά δεύτερον θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρωση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές σε σχέση με το FC. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Και αυτό θεωρώ ότι εξηγεί τι αλλαγέ που έγιναν στα θέματα κυβέρνηση. Φυσικά και ακούσαμε κάποια κρατική, η οποία ενδεχομένω ε, να πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιες αλλαγές στη φάση των πραγματεύσεων και θα κοιτάξουμε και τα σχόλια των άλλων επιτροπών, των καθήλια αρμόδιων επιτροπών. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο δυναμικό για αλλαγές. Αλλά πιστεύουμε ότι θα ήταν λάθος να γίνει απλά μια σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση με το ΕΦΣΥ γιατί είναι διαφορετικό πολύ απλά το εργαλείο και είναι διαφορετική κατάσταση. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. για τα θέματα τα οποία ακούσαμε. Να κάνω κάποια σχόλια στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι πολλά ακούσαμε για τα θέματα των προτεραιοτήτων. Κατανοήσουμε προφανώ το γεγονό ότι καταλαβαίνουμε ότι η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή σα είναι πιο πολύ εστιασμένη στο άρθρο 2. Να τονίσω αυτά που ακούσαμε, ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προβολή σε ό,τι αφορά το τι σημαίνει το παράδειγμα 2 για τις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων και αυτό θα το μοιραστούμε σύντομα με την Επιτροπή σας. Και νομίζω ότι πιο πολλές τροπολογίες μπορούν είτε να συμπεριληφθούν στην ε, βασική πράξη και πολλέ και στις κατευθυντήριε γραμμές για τις επενδύσεων γιατί έχουν να κάνουν με τις προτεραιότητες. Συνολικά καλωσορίζουμε τις προτάσεις που γίνονται και σε άλλους τομείς σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Και υποστηρίζουμε την ιδέα του InvestEU να προωθήσει τους στόχους του TNT, αλλά και τις οριζόντιες προτεραιότητες, όπως η μείωση της, του άνθρακα, σε ό,τι αφορά τις ανακτικές μορφές ε, μεταφορών. Άρα, Φανταζόμαστε ότι μεγάλο τμήμα των τροπολογιών θα αποτυπωθεί στι κατευθύνσει γραμμέ για τι επενδύσει. Το θέμα τη κλιματική αλλαγή, από ό,τι κατάλαβα, προκαλεί κάποιε ανησυχίε. Και ενδεχομένω να το δούμε και από μια διαφορετική γωνία. Κατανοούμε τι ανησυχίε σα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η DG Move υποστηρίζουν ένα φιλόδοξο στόχο. Σύμφωνα και με αυτά που αποφασίσαμε στο Connecting Europe Facility. Πρέπει να συζητήσουμε τώρα το επίπεδο του στόχου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια για το πώς θα προσμετρηθεί αυτός ο στόχος. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουμε και άλλους τομείς, άλλους τρόπους μεταφορών και όλοι αυτοί οι τρόποι μεταφορών θα πρέπει να καταμετρηθούν με κάποιο τρόπο για να δούμε τι σημαίνει αυτό για την αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, συνεκτικός τρόπος λοιπόν ε, προσμέτρησης της επιτευξής των στόχων και πιστεύουμε ότι ο στόχος του καθεαυτός μπορεί να επιτευχθεί. Το θέμα το οποίο έφερε συνάδελφος, δεν θα το αναλύσω εγώ. Αυτά. Σας ευχαριστώ από την κυρία, από την DG Τώρα το λόγο να πάρει ο κ. Βίντε Φανελκάμπ για να ολοκληρώσω τη συζήτηση για να συνοψίσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τρει παρατηρήσει έχω να κάνω. Τέσσερι, μάλλον. Καταρχά, η συντήρηση, το maintenance, δεν είναι αρμοδιότητα του EU Invest. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει, έχω εξ αρχή. Μιλάμε για νέε επενδύσει και τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, έργα υποδημών είναι τα ίδια αρμόδια για τη συντήρηση. Δεύτερη παρατηρήση σε ό,τι αφορά τους κλιματικούς στόχους. Και την κυρία Κριστίν να την παραπέμψω στην γνωμοδότηση της 28ης Μαρτίου 2018. 17, συγγνώμη, για το ΕΦΣΙ, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει στόχος 40% χρηματοδότησης από το ΕΦΣΕ. 30, 40, 50. Ρε και κυρία Κριστίν και Κοσμά, νομίζω ότι στο 40% είναι η χρυσή Είναι φυσικά μεγάλος ο διαλυσμός σας, αλλά η πραγματικότητα πολύ απλά είναι διαφορετική. Η κερδοφορία τώρα. Κοιτάξτε, με τον σεβασμό που θα τρέφω είναι μάλλον κομμουνιστική αυτή η αντίληψη φυσικά και χρειάζεται να υπάρχει κέρδος. Όταν ε, ένας εργολάβος αναλαμβάνει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό έργο, τι το αναλαμβάνει άμα είναι να μην βγάλει κέρδος. Τι να πάμε δηλαδή πριν από την ε, Γαλλική Επανάσταση σε τέτοιες εποχές. Τώρα πρόεδρε για θέματα διακυβέρνησης. Δεν συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέει, ότι θέλει πιο πολύ να χαράξει πολιτική. Σύμφωνοι. Γιατί θέλουμε πιο πολύ πράσινη προσέγγιση, θέλουμε καινοτομική προσέγγιση, αλλά εδώ μιλάμε για δάνεια. Τα δάνεια αυτά πρέπει να έχουν και σύμφωνα με το ΕΦΣΙ μια κάποια αξία στην αγορά. Οι επιδοτήσει είναι στο ΣΕΦ. σε άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τι επιδοτήσει. Τα εμπορικά όμω, δάνεια, οι εμπορικέ πιστώσει, θα τι ε, επιμολύνουμε εισαγωγικά με πολιτική. Αυτό είναι πολύ αμφισβητήσιμο. Μπορούμε να πούμε και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρχει πολυτροπικότητα στι μεταφορέ, διασυνοριακότητα, πράσινη προσέγγιση. Σύμφωνοι αλλά τον αναλάβουμε εμείς την διακυβέρνηση, γιατί θέλουμε να βάλουμε πιο πολιτικούς στόχους, δεν ξέρουμε πώς χάσουμε τελικά και τα δάνεια τα ίδια. Αυτό θα το συζητήσουμε στη συνάντηση των σκιωδών μαζί με την Σύμβολη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και Ευχαριστούμε τον κύριο Βίμ Φαντενκάμπ και να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος μην Φαντεκάμπ μπορεί να είναι τοπικά αυτά τα οποία διακηρύττω, αλλά χωρίς ε, αυτή την τοπία δεν υπάρχει καμία γόνιμότητα σε ό,τι αφορά τις δράσεις μας. Χρειάζεται λοιπόν και αυτός ο τοπικός χαρακτήρας όταν μιλάμε για θέματα κλίματος. <laughs> Και να σας υπενθυμίσω ότι η έκταση του κυρίου Βινφανεκάμπ για κατασταση τροπολογιών 5η 27 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα η προθεσμία. Και συνεχίζουμε, αλλά πριν το μικρόφωνο της Πρόεδρου. Madame Messner n'est pas encore là et donc je vais suspendre notre séance. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 15 λεπτών, γιατί η συγγήτρια για το επόμενο θέμα δεν έχει έρθει ακόμα. 15 λεπτά. Κύριε Δαβενταλόν, μήπως είναι εδώ όλοι οι βουλευτές που θέλουν να συζητήσουν την έκθεση που είχαμε προγραμματίσει για τις 6 το απόγευμα, δηλαδή για την πρόταση κανονισμού για τα ε, Μία περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής. Το ΕΛΚ είναι εδώ, ναι, το ECR, ναι, ο κύριος Λατόφσκι. Για την άλλη δεν είναι εδώ. Ο κύριος Ρικέ. Συγγνώμη κύριε Ρικέ, σας ε, ξεχνάω σήμερα. Περίεργα πράγματα. Πρώτες τις χειρές Νταλών, λοιπόν, μήπως να συζητήσουμε τώρα αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Συμφωνείτε? Ωραία. Εντάξει, για να μην κάνουμε και διάλειμμα άσκοπα. Ωραία. Θα περάσουμε λοιπόν στο σημείο 8 και μετά θα γυρίσουμε στο 6 της κυρία ε, Κυρία Ρεβονταλόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, συνδέεται αυτό που θέλω να σας παρουσιάσω με την προηγούμενη έκθεση. Πρόκειται για την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας σε σχέση με τις προτεραιότητες του Ταμείου Συνοχής και του, Ταμείου, ε, του Περιφερειακού Ταμείου. Μας δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην καθορισμό των προτεραιοτήτων. Θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει πολλά προβλήματα, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη της ε, ότι οι περιφέρειες μπορούν να αξιοποιούν το εργαλείο της συγχρηματοδότησης δεν έχει στο στρατηγικό στόχο ΣΕΦ ε, ε, δεν έχει μάλλον συμπεριλάβει την λεγόμενη ε, θεματική προσέγγιση στον τρίτο στόχο, το ΣΕΦ. Για το στρατηγικό στόχο 1 το κάνει το ίδιο και για τον δύο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε συγχρηματοδότηση υποδομών για τις μεταφορές. Προτείνω λοιπόν. Το πέρασμα. Να υπάρξει μια ε, χρήση των διαθέσιμων πόρων και για την χρηματοδότηση προγραμμάτων υποδομών για τις μετηφοράς πρόσφυγε συγκεκριμένα 25% για τις περιοχές που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο και 20% για τις ε, ε, πιο αναπτυγμένες περιφέρειες. Θεωρώ επίσης ότι δεν είναι λάθος να μην έχουμε αντίστοιχες ε, δυνατότητες για εκείνες τις, τις, τις πιο αναπτυγμένες περιοχές. Προσπαθώ λοιπόν με την γνωμοδότησή μου να προτείνω διορθώσεις, ε, ειδικά σχετικά με τις μεταφορές, πρώτα απ' όλα για τις έξυπνες μεταφορές και τη δυνατότητα να προωθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τον στρατηγικό στόχο της ευφιέστερης Ευρώπης. Μετά, να αξιοποιηθούν αντίστοιχοι πόροι και για τον στόχο του στρατηγικό 2. Οι μεταφορές είναι και αυτές ένα εργαλείο για την ε, μεγαλύτερη περιφερειακή συνοχή, επομένως μπορεί να ταιριάξει και με το στρατηγικό στόχο 3 και επίσης με τον 4 γιατί μιλούμε για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Και άρα δηλαδή τον στρατηγικό στόχο για την καταπολέμηση των κοινωνικών αποκλεισμών στην Ευρώπη. θέλαμε λοιπόν να μπορούν να επωφεληθούν από αυτά τα ταμεία και ε, τα, οι, περιφέρειες έτσι ώστε να, να, ε, βελτιώσουν τα αεροδρόμια τους ή το τροχαίο υλικό των σιδηροδρόμων τους. Κύριε Φαντεμπκάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω την τιμή σήμερα το απόγευμα να αντικαθιστώ την αγαπητή συνάδελφο Κλάουντα Μοντέρο Αγγίλα η οποία είναι ακόμα ε, σε άντια, μητρότητος. Σας στέλνει χαιρετίσματα. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για την προσέγγιση της, αλλά είμαι λίγο πιο προσεκτικός και επιφυλακτικός από ότι η εισηγήτρια. Πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με διάφορες τέτοιες ε, αρμοδιότητε και διάφορα τέτοια καθήκοντα. Πρόκειται για ένα ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη, Όσο πιο πολύ μεταφορά μπορούμε να βάλουμε και όσο πιο καινοτομικό και πράσινο είναι ο τρόπο που μπορούμε να βάλουμε τέτοια ζητήματα, τόσο καλύτερο. Αλλά να μην, υπο, να μην υποτιμούμε την Επιτροπή Μεταφορών για το DRD. Αποτελεί τμήμα τη όλη συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικού πλαίσιο και έχουμε πρόσφατα εγκρίνει και την έκθεση του κυρίου Ρικέ, την γνωμοδότηση μάλλον προς την Επιτροπή Προπολογισμού για το πώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημορφωθεί αυτή η ισορροπία και αφαιρείται ένα μεγάλο ποσό από το ERDF υπέρ του ΣΕΦ. Αν λοιπόν η Κριστίν ε, επιβαρύνει το ERDF μήπως τελικά αναλαμβάνουμε υπερβολικά μεγάλες αρμοδιότητες, άρα η σχέση μεταξύ πουδουπού ταμείων συνοχής και ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης, όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν, να, να λειτουργούν με μια καλή ισορροπία. Ένα μεγάλο πρόβλημα για το ΕΛΚ λοιπόν είναι η περικοπή επενδύσεων σε αρρολιμένες στις εξόχως από κεντρές περιοχές. Εδώ θα πρέπει να επιτύξουμε μεγάλη προσοχή, πιστεύουμε. Γιατί πολλά εξαρτώνται από αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολλά αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια σε ρυθμό, όχι όμως τις απόκεντρες περιοχές και θα θεωρούσαμε ότι θα ήταν μεγάλο κρίμα να υπονομευθούν αυτά τα έργα. Θα κάνουμε λοιπόν επικοδομητικές τροπολογίες προκειμένου να είναι καλή η έκβαση της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει και η πρόεδρος, η κυρία Στουλόσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότηση. Η πολιτική συνοχή είναι η πιο σημαντική πηγή χρηματοδότηση των σχεδίων των έργων υποδομών και το μόνο εργαλείο που μα επιτρέπει να συμπεριλάβουμε τι πιο φτωχέ περιοχέ στο δίκτυο ευρωπαϊκών μεταφορών ε, και να γίνει αυτό ένα δίκτυο συνοχή. Γι' αυτό η υποστήριξη των υποδομών σε όλου του ε, τρόπου μεταφορών θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με σήμερα. Θα πρέπει να κρατήσουμε επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επενδύσεων και στα αεροδρόμια, ας πούμε, και στην αγορά ε, συνδρομικού υλικού. Η Κομισιόν πρότεινε να αποκλείσουμε το συνδρομικό τομέα. Αυτό είναι φραγμός για τις ε, πολύτροπες μεταφορές. Ε, θα είναι εμπόδιο και για να περιορίσουμε τις ε, εκπομπές διοξιδίων από, τα, τις χερσιές μεταφορές. Ε, νομίζουμε ότι είναι μια εναλλακτική ένας εναλλακτικός ε, τρόπος μεταφοράς φορτίου και επιβατών σε σχέση με τις χερσαίες μεταφορές. Επίσης, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχουμε όλο και περισσότερες ανάγκες. Και μια και η αγορά και ο αριθμός των επιβατών αυξάνεται, και ναι, μεν στο παρελθόν είχαμε προβλήματα αποτελεσματικότητα στι εναέριε μεταφορέ, αλλά στην Πολωνία τουλάχιστον κάθε χρόνο τα τοπικά αεροδρόμια εξυπηρετούν το και περισσότερου επιβάτε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν με το να αποκλείσουμε τα περιφερειακά αεροδρόμια από τη χρηματοδότηση των, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι κρίμα. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τους κλιματικούς στόχους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, προβλέπει ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση αυτή για το κλίμα να είναι 30%. Ε, όμως ε, υπάρχει ένα κατόφλι του 37% και το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο μας λέει ότι θα πρέπει τουλάχιστον να είναι το 25% του κοινοτικού προϋπολογισμού που θα πρέπει να δαπανάτε για να υλοποιήσουμε τους κλιματικούς στόχους. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί, πιο ευέλικτοι για να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες και τις, την πραγματικότητα των διαφορών κρατών μελών. Το επίπεδο θεματικής συγκέντρωσης θα πρέπει να καθοριστεί σε διάλογο με τα κράτη-μέλη, με τρόπο εξατομικευμένο για να εντοπίσουμε καλύτερα τα στοιχεία όπου πρέπει να στήριξουμε περισσότερο. Ε, η πρόταση θεματικής συγκέντρωσης. Ε, για αυτή την πρόταση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολύ συχνά η περιφέρεια σε ένα κράτος μέλος δεν, ε, χρησιμοποιούν τόσο καλά τα ευρωπαϊκά κονδύλια όσο Σε εθνικό επίπεδο όμω μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα του φραγμού και να καταστήσουμε αυτή τη διαδικασία πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να δώσει θετικά στοιχεία η διάγνωση και οι λύσει τη Κομισιόν ε, μα φαίνονται δικαιολογημένε. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότηση, είμαστε ικανοποιημένοι με τη γενική κατεύθυνσή του. Συμφωνούμε με πάρα πολλά σχόλια, ειδικά αυτά που αφορούν την ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και την πολιτική συνοχή. Φυσικά θα καταθέσουμε τροπολογίες και βασιζόμαστε στην καλή συνεργασία στα πλαίσια των ε, του διαλόγου που γίνεται με τους σκιώδεις εισηγητών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρικία έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαίρω την Κριστίν για την επινοητικότητά της, την ευρηματικότητά της, την ικανότητά της να ανανεώνει το περιεχόμενο της έκθεσης, μια γενική παρατήρηση ε, που θα καλύψει όλα όσα άκουσα και από την εισηγήτρια και από τον Βιμ Βαντενκάμπ και από τον κύριο Σλοτόφσκι. Το πρόβλημα για μας, την, την Επιτροπή δηλαδή Μεταφορών, είναι ότι τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, δεν πηγαίνουν προς τις μεταφορές που μας, θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς, με προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ένωσης, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό είναι και θεματικό και γεωγραφικό θέμα. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω και το είπε και ο κ. Λουτόφσκι μόλις τώρα, είναι ότι σε περιφερειακό επίπεδο συχνά δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε αυτά τα ταμεία, ε, τα κονδύλια από τα ταμεία, ε, γιατί τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι πάρα πολύ δεσμευτικά με πολλούς περιορισμούς. Συμπέρασμα, συχνά καθυστερούμε. Ειδικά τα πρώτα χρόνια υπάρχουν πολλά προβλήματα και η κατανάλωση των περιφερειακών κονδυλίων δεν είναι βέλτιστη. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι και σε θεματικό επίπεδο, δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά τη χρήση των κονδυλίων και την ευκολία χρήση του και στον τρόπο κατανάλωση. Ακριβώ γι' αυτό θα πρότεινα στα πλαίσια αυτή τη πρόταση τη Κομισιόν, κάτι που πρότεινα και σε άλλε επιτροπέ, είναι να μεταφέρουμε 20 δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη για την Ανταγωνιστικότητα προ το μηχανισμό διασυνδέοντα την Ευρώπη. Κάτι που καλύπτει όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Θα μας εξασφαλίσει όλα αυτά που θέλουμε. Δηλαδή και θα πάει ε, προς μια κατεύθυνση θεματικά ικανοποιητική και θα δώσουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσα από αυτά τα θέματα. Θα υπάρχει μεγάλη απλούστευση σε επίπεδο κρατών μελών και είμαστε σίγουροι ότι η κατανάλωση θα είναι σωστή γιατί όπως ξέρετε ο μηχανισμός ε, είχε πολύ συμμετοχή, κάτι που δεν συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά ταμεία. Επίσης, επί της ουσίας, τα, τα ταμεία συνοχής ήταν ε, σημαντικά για, την, για τις χώρες συνοχής ε, μέσω αυτής της μεταφοράς αυτών των 20 δισεκατομμυρίων. Παλιά ήταν 10 δισεκατομμύρια από τα 80, έτσι. Ίσως τώρα έχουμε φτάσει, μπορούμε να φτάσουμε σε 45%. Είναι πολύ σημαντικό, ε, και το 20% του Ταμείου Συνοχής. Ε, εδώ προτείνω 20 δισεκατομμύρια, έτσι, ε, σε σχέση με τα 320 δις. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να περάσει. Δεν θα φτάσει όμως, ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει με μέχρι τον προπολογισμό και να υιοθετηθεί τελικά, αν δεν περάσει από όλε τι επιτροπέ. Νομίζω ότι θα εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή προστατευμένη αξία και αποτελεσματικότητα και απλότητα. Και νομίζω ότι και το Συμβούλιο θα τη θέλει. Γιατί επιτρέπει να δώσουμε στα κράτη ε, μία δυνατότητα να προωθήσουν προγράμματα κοινού ενδιαφέροντο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ε, να ανταποκριθούμε στους στόχους με το να ορίσουμε νέους ε, στόχους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Γιατί μπορούμε να κάνουμε καλύτερο προσανατολισμό προς στόχους για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, συχνά είχαμε δυσκολίες να προωθήσουμε προγράμματα που είχαν σημαντική ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και είχαν και δυσκολίες οι περιφέρειες. Γιατί η ανάγνωση των προγραμμάτων, η ερμηνεία των προγραμμάτων και το γεγονός ότι οι περιφέρειες ε, θα έπρεπε να προωθήσουν αυτά τα προγράμματα, ε, τις δυσκόλευε θα πρέπει να δούμε το βαθμό ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας. Μερικές φορές ε, αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα ήταν πολύ συγκεντρωτικά, ε, ήταν δύσκολο να τα διαχειριστούν οι περιφέρειες. Και μια, έτσι ένα προβληματισμό. Καταλαβαίνω την ε, Κριστίν, ε, η οποία έχει, την ενδιαφέρει πολύ το κοινωνικό θέμα. Θέλει να επαναπαρασοανατολίσει, να δώσει έμφαση μεγαλύτερα το πιθανό κοινωνικό χαρακτήρια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακή Ανάπτυξη. μην ξεχνάμε όμω και το κοινωνικό ταμείο. Δεν το συζητάμε σήμερα. Ξέρω ότι έχει άλλη φύση χρηματοδότηση του ενό ταμείου σε σχέση με το άλλο, αλλά πρέπει να υπάρξει μια διασύνδεση ανάμεσα στα δύο ταμεία. Να το ξαναδούμε αυτό παρά να δώσουμε μεγαλύτερο κοινωνικό χαρακτήρα σε αυτές τις πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πάντω, η έκθεση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί πάει στην ουσία, στο, στο ψητό και προσπαθεί να περάσει και να προωθήσει νέους στόχου με συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις, λοιπόν, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, λοιπόν, Χριστίν. Ευχαριστώ, κύριε Ρικέ. Ο κύριο Τέιλορ έχει το λόγο. Ε, um, um, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μέρο του κυρίου Evans. Τη κυρία Evans. Μιλώ. Πιστεύει ότι οι επενδύσεις στα έργα υποδομής για τις μεταφορές θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Ελαχιστοποιώντα και το κόστος βεβαίως. Αυτό αυτή η έμφαση, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να ε, είναι ξεκάθαρη και όταν ε, το χρηματοδοτούμε περιφερειακά αεροδρόμια. Όταν για παράδειγμα έχουμε δύο ξεχωριστά περιφερειακά αεροδρόμια στις δύο πλευρές ενός συνόρου. Ε, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας για παράδειγμα. Και εάν πράγματι θέλουμε να φροντίσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να δούμε τέτοια και να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Δεν ε, είναι αυτό απλώς ένα ζήτημα ε, ποια περιφέρεια, ποια περιοχή θα, έχει μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές. Όλοι ζούμε στην ίδια περιφέρεια που ονομάζεται πλανήτης Γη. Αυτά τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικές συγχρηματοδοτούμενες από το Connecting Europe. Για τη δημιουργία λέγεται υποδομών ε, όπως γέφυρες, όπως αυτοκινητόδρομοι και τα υπόλοιπα να χρησιμοποιηθούν για άλλα προγράμματα όπως για παράδειγμα μείωση του θορύβου ή ε, την ε, ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρόμων στο ΕΤΕΝΤΗ. Έτσι λοιπόν προτείνουμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτό και έτσι θα συνεισφέρουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρικέ, κύριε Δεμόντε, έχετε ζητήσει το λόγο. Συμφωνώ με την Κριστίν. Ως προς το ότι τα, τα μία για τα οποία συζητούμε, η πρώτη τους προτεραιότητα θα πρέπει να είναι, η, μάλλον οι προτεραιότητες θα πρέπει να πηγάζουν από τις περιφέρειες. Θα πρέπει οι περιφέρειες να θέτουν τις προτεραιότητες στη χρήση αυτών των χρημάτων. Γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι ίσως υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις μεταφορές και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των ανταλλαγών και των σχέσεων μεταξύ των διαφέρων περιφερειών. Υπάρχουν ίσως κάποιοι τομείς στους οποίους να υπάρχουν επικαλύψεις. Ε, Όμω αυτό δεν είναι ένα αναγκαστικά πρόβλημα. Μπορούμε για παράδειγμα να υποστηρίξουμε τον ε, τουρισμό. Έχουμε ήδη συζητήσει και έχουμε ήδη ακούσει σε αυτή την Επιτροπή ότι αναμένεται μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των επιβατών μέχρι το 2050. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί απλώς αυξάνοντας τη χωρητικότητα των αεροδρομίων, γιατί το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να έχουμε μεγάλα ποτηλιαρίσματα στους δρόμους γύρω από τα αεροδρόμια. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε άλλους τρόπους βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών. Επίση, όσον αφορά τι απόκεντρε ή εξόχω απόκεντρες περιφέρειες. Αυτές τις περιφέρειες θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε ιδιαίτερα ε, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη και καλύτερη σύνδεση με τις υπόλοιπε περιοχέ, με τις υπόλοιπε περιφέρειες. Και θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο, στα παραρτήματα υπάρχει ο μαθηματικός τύπος για να υπολογιστεί η συγχρηματοδότηση, το άρθρο 9 συγκεκριμένα. Στην σελίδα 179. Εδώ αναφερόμαστε σε, εξόχο, σε απόκεντρες περιοχές και σε ε, περιοχές ε, διασυνοριακές, με, με, δύο πλευρές ενός συνόρου θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξή. Όταν θα κάνουμε, όταν θα υπολογίζουμε το, τα, βάρη σε αυτόν τον τύπο, θα, θα κοιτούμε το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε, σε μια ακτίνα 25 χιλιόμετρων, σωστά το έχω καταλάβει. θα ήθελα να εξηγήσετε ποιε είναι οι επιπτώσει αυτού του τρόπου υπολογισμού για τι εξόχω απόγεντρε περιοχέ. Γιατί αν το έχω καταλάβει σωστά, έχω την εντύπωση ότι κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υποστηρίζει τις ε, περιφέρειες τις ε, πιο απομακρυσμένες της. Αντιθέτως, φαίνεται σαν με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού να οδηγούμαστε σε μια μεγαλύτερη ενίσχυση των αστικών περιοχών. Να δώσουμε μέσα λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you very much, Chair, and thank you for the opportunity um, to... Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Επιτροπή σας. Να ξεκινήσω καλωσορίζοντα το σχέδιο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και κυρίω για την ταχύτητα με την οποία εργάστηκε. Γιατί, όπω είπαμε, πρόκειται για μία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι οποίε έχει τονίσει η Πανελλημένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ανάγκη να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε όλο το πακέτο του Πουδουπού. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να επανέλθω στην τελευταία ερώτηση. Αν σωστά κατάλαβα την ερώτηση, νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με τα παρατήματα του κανονισμού των κοινών κανονισμού γενικών διατάξεων. Προτεραιότητα υποστηρίξης, λοιπόν, για, τις πολιτικές, ε, για την πολιτική συνοχή, για την συνοχή, παραμένει οι πιο αποκεντρωμένες περιοχές και μάλιστα η πρόσθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυξάνει το ποσό χρηματοδότηση σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο για τις πιο απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. Δύο σημεία επιτρέψτε μου να σχολιάσω. Καταρχάς το θέμα της θεματικής συγκέντρωσης και το τι προσπαθεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη χρήση των Ταμείων Συνοχής και των Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της θεματικής επικέντρωσης. Να σας το πω απλά. Ο σκοπός της θεματικής επικέντρωσης είναι να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες της Ένωσης με έναν ανάλογο βαθμό φυσικά ευελιξίας προκειμένου οι περιφέρειες να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις ε, ανάγκες τους. Κάποιες ε, από τις ε, προτάσεις στη θεματική επικέντρωση μας παρουσιάζουν προβλήματα. Καταρχάς, επεκτείνοντας την ιδέα της θεματικής επικέντρωσης στους τρεις από τους πέντε στόχους προτεραιότητα, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για επικέντρωση, γιατί αν μιλάμε για τρεις από τις πέντε προτεραιότητες πώς μπορούμε να μιλήσουμε για βασική προτεραιότητα και συμπληρωματικά, κοιτώντας και τα αριθμητικά στοιχεία που προτείνονται. Ο βαθμός θεματικής επικέντρωσης έτσι όπως αναλώνεται στις τρεις προτεραιότητες, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση, θα απαιτούσε μεγαλύτερο βαθμό θεματικής επικέντρωσης σε σχέση με αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι αντίθετο με αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Με την ευελιξία που είπαμε ότι χρειάζονται οι περιφέρειες για να προσαρμόσουν τη χρηματοδότηση στις ανάγκες τους. Αυτό έχει να κάνει και με το λόγο για τον οποίο ε, προτείνουμε θεματική επικέντρωση σε εθνικό επίπεδο και όχι σε περιφερειακό επίπεδο ο συνήθω. Κάποιοι μίλησαν για μια ενδεχόμενη κεντρική διαμόρφωση της διαδικασίας. Για να υπάρχει ε, έλεγχο σε επίπεδο πρωτεύουσών και όχι τόσο πολύ περιφέρειε. Αλλά ο σκοπός μας είναι ο αντίθετο. Τη στιγμή έχουν, που υπάρχει η περιφερειακή επικέντρωση, σε περιφερειακό επίπεδο ορίζονται και τα ποσοστά, ενώ όταν υπάρχει επικέντρωση σε εθνικό επίπεδο, τα ποσά σε περιφερειακό επίπεδο είναι ευέλικτα. Εφόσον φυσικά τηρείται το εθνικό όριο. Δύο τελικά τελευταία σημεία επιτρέψτε μου να κάνω, να σχολιάσω. Ακούσαμε δύο λόγια για την επικέντρωση σε στόχους κλιματικούς. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε τους λόγους που μας οδήγησαν στα ποσοστά που προτείνουμε. Προτείνουμε 25% γενική προσέγγιση, 25% σε ό,τι αφορά τον ε, προπολογισμό μετά από το 2020 για τους κλιματικούς στόχους. Και ένας βουλευτής είπε ότι τα ποσά που προβλέπονται για τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής είναι πιο υψηλά. Αυτό είναι σωστό και έγινε σκούπιμα, γιατί κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει αυτό που τον αλογεί. Προφανώς και τα μία αυτά μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στον, στην επιτεύξη των στόχων των κλιματικών. Ενώ, για παράδειγμα, άλλα, άλλα ταμεία μπορεί να έχουν πρόβλημα να πετύχουν το 25% όπως το, για παράδειγμα το Ταμείο Συνοχής. Ένα τελικό τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσει που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ένα βουλευτή εξέφρασε σχετικέ ανησυχίε. Να τονίσω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με κάποιε από τις εξαιρεσει είναι να εξαγάγουμε δύο, αν θέλετε, διδάγματα από το παρελθόν. Να υπάρχει καταρχάς ε, γουργός χαρακτήρας σε ό,τι αφορά αυτά που είδαμε και στο παρελθόν και να υπάρχει και συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εξαίρεση των αεροπορικών υποδομών. Σύμφωνα και με την έκθεση του Ρεκτικού Συνεδρίου πριν από 2-3 χρόνια που ήταν πολύ αρνητικό για τη χρηματοδότηση περιφερειακών αεροδρομίων και πιστεύουμε ότι αυτό καλύτερα να μείνει στα χέρια των εθνικών αρμοδιοτήτων, να υπάρχει δηλαδή εκεί η πρόβλεψη για τη σωστή χρηματοδότηση. Και τέλος, ε, για το τροχαίο υλικό. Θα πρέπει να φροντίσουν οι εταιρείε τελικά. Να μην υπάρξει υπερβολική και άδικη επιβάρυνση των επιβατών. Ευχαριστούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και με τους Χιώδες και με τα υπόλοιπα μέλη και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Προσβλέπω λοιπόν σε αυτή την υποκοδομητική συνεργασία που θα έχουμε. Πάντως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, να, να αναγνωρίσουμε ότι οι μεταφορές είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους και όταν αναφέρομαι στην κοινωνική διάσταση, Ντομινίκ, αναφέραμε ακριβώ το γεγονό ότι οι μεταφορέ, το να έχει κανεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο μεταφορών, μπορεί να καταπολεμήσει τον αποκλεισμό τη μια περιφέρειας και βοηθάει στι ανταλλαγέ μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Γι' αυτό λοιπόν οι μεταφορέ είναι ένα θεμελιώδου σημασία άξονα και που, το οποίο θα πρέπει να τον προωθήσουμε και στο ε, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και, στο, και σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο ή ε, νομοθετικό εργαλείο συζητούμε. Ε, είναι σημαντικό όμως να λαμβάνουμε υπόψη να τις μεταφράσει όχι μόνο για ορισμένους στόχους αλλά για όλους τους στόχους και ακόμη περισσότερο να βοηθήσουμε εκείνες τις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αυτές που είναι πιο απομακρυσμένες για παράδειγμα ή που είναι λιγότερο αναπτυγμένες. Αλλά και τι άλλε, τις περισσότερο αναπτυγμένες, θα πρέπει να δούμε τους στόχους, έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική προσέγγιση και προσεκτική. Για να χρηματοδοτήσουμε εκείνα τα έργα ε, που θα έχουν τελικά αποτέλεσμα από την πλευρά των περιφερειών γιατί βεβαίω υπάρχει και το επίπεδο των κρατών μελών, αλλά εμεί εδώ πιστεύω ότι κάνουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολύ αποτελεσματική, έχουμε μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία με τι περιφέρειε. Και τελικά σε ορισμένε περιπτώσει, μάλιστα ορισμένε περιφέρειε καταφέρνουν να προχωρούν και να προοδεύουν καλύτερα και από το κράτο μέλου του. Εκεί πρέπει να τι βοηθήσουμε. Σα ευχαριστώ. Αυτέ τι παρατηρήσει είχα να κάνω Δεν χρειάζεται να με λέτε Μαντάμ Χριστίνη, θα λέτε όλο μου το επώνυμο, ή θα λέτε Χριστίν. Γιατί τους άντρες ε, βουλευτές ξέρετε να τους ε, ονομάσετε. Ευχαριστούμε κυρία Βονταλόν και για το μικρό σας όνομα. Δεν αποκαλούμε τους συναδέλφους ε, με το μικρό τους, έτσι, αλλά με το επώνυμο. Και σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις επί της έκθεσης που, δίνει τη σχέση, που δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην Ευρώπη και στα εδάφη μας. Γιατί χωρίς τα εδάφη μας δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την Ευρώπη. Ε, υπενθυμίζω ότι Δευτέρα 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι έχει την προθεσμία για να καταθέσετε τροπολογίες. Πάμε στο σημείο 6. Κυρία Γεζίν Μέσνερ είναι εδώ. Λοιπόν, χωρίς ανάσα, πάμε στην πρόταση οδηγίας ε, για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, ε, παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων αποβλία. Ε, θα καταργηθεί η οδηγία 2009-16 και θα... Συγγνώμη, θα καταργηθεί η οδηγία 59 και θα τροποποιηθεί η οδηγία 2009-16 και η οδηγία 2010-65. Η κυρία Μέσνα έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που αλλάξατε την ε, ημερήσια διατάξη, γιατί ήθελα να ψηφίσω στην Επιτροπή Ήτρε που είχα ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε ιδιαίτερα. Και τώρα πλέον ε, είμαι έτοιμη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, τις λιμανικές εγκαταστάσεις παραλαβής έχουμε ήδη οργανώσει μια συνάντηση των σκιωδών. Πήγε καλά κάναμε ανταλλαγή απόψεων και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε Πώ αξιολογούν κάποιες αλλαγές που θέλαμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να πούμε ότι γενικώ πώς ε, κάναμε λίγο πιο έντονη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε. Να σας πω ότι και την πρώτη πρόταση θεωρού, τη θεώρησα καλή. Αυτή την ε, προσέγγιση λοιπόν σε ό,τι αφορά την ε, μία ενιαία λύση για όλους τους λιμένες. Ε, είχα τις αμφιβολίες μου γιατί εξέτασα και την κατάσταση στην Γερμανία, την Ολλανδία, τη Λισαβόνα και σε άλλες χώρες και διαπιστώσα ότι πραγματικά θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις γιατί πρόκειται για οδηγία. Η οδηγία σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο προσαρμογής από πλευρά του κράτους μέλους αλλά θέλουμε να δούμε τι είναι πραγματικά εφικτό. Και αυτό κάναμε και στην συνάντηση των σκιωδών. Αύριο λοιπόν θα συνειδηθούμε εκ νέου με, τον, με τους σκιώδες και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε μία ενιαία έκθεση, να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία. Έχουμε ως τώρα 8 συμβαστικές προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά το παιδί εφαρμογής. Καταρχάς δεν αλλάξαμε και πάρα πολλά εδώ. Βάλαμε το reasonable και practicable, δεν είναι και μεγάλη διαφορά. Στο άρθρο 4, σε ό,τι αφορά τις άμεσες ε, λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, ε, θέλουμε να τονίσουμε ότι θα επικεντρωθούμε και στα θέματα ανακύκλωσης. Να χρησιμοποιηθεί και η έντζα. Ξέρω ότι αυτό δεν το έχει κατά νου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευθύ εξ αρχή μεταβήκαμε με μια μικρή αποστολή στην ΕΜΖΑ και ανάφερε η ΕΜΖΑ ότι διαρκώ αποκτά νέε αρμοδιότητε, αλλά όχι καινούριου πόρου και καινούριο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί ε, από την αρχή του προγράμματο η ΕΜΖΑ. Έχουμε και τις ε, εξόχους κεντρικές περιοχές, οι οποίες και αυτές συμπεριλήφθησαν. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις ε, τοπικές ιδιαιτερότητες τους να χρησιμοποιούν ε, ανάλογα κονδύλια γιατί φυσικά αλλιώς τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ στην Ευρώπη. Ύστερα, σε ό,τι αφορά τις μονομένες εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, είπαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια κατανομή των πληροφοριών σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη δομή του κόστους ε, εδώ τονίζουμε ως κοινοβούλιο ότι τα αγγλικά είναι σημαντική γλώσσα γιατί αποτελεί την κοινή γλώσσα, τη διεθνή γλώσσα επικοινωνίας. Διευκρινίσαμε λοιπόν το τι πληροφορίε πραγματικά χρειάζονται για να ξέρουμε που βρισκόμαστε και τα θα πρέπει να είναι σαφές επιπία βάση υπολογίζονται τα τέλη τα οποία καλύτερα να υποβάλει, να καταβάλει κανεί. Και ότι σε ό,τι αφορά του μικρού λιμένε, μπορεί να υπάρξει συνεργασία. Αυτό μα απασχολεί ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τώρα την επιπτία την οποία θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνεται κάθε τρία χρόνια, Εμεί θέλουμε να γίνει κάθε πέντε χρόνια. Σε μικρού λιμένε, λοιπόν δημιουργήσαμε διάφορε προποθέσει για την εξαίρεση, για παράδειγμα των μικρών λιμένων, εάν συμμετέχουν στο περιφερειακό σύστημα και αν αυτό μπορούν να το αποδείξουν και αν το αναφέρουν αυτά τα κράτη-μέλη δεν θέλουμε να μη συμπεριλαμβάνονται οποιασδήποτε εγκαταστάσεις αποβλήτων. Σε ό,τι αφορά την άμεση μεταφορά των αποβλήτων από το πλοίο τώρα. Φυσικά δεν μπορούν αυτά τα απόβλητα να απορρίπτονται στη θάλασσα. είναι σημαντικό να το βάλουμε αυτό. Ξεκάθαρα. Και το σχέδιο για την παράδοση αποβλήτων ήταν σημαντικό να αναφερθεί αυτό στους μικρούς ε, λιμένες. Ε, αναφέραμε διάφορες ε, ιδιαιτερότητες και κάποιοι είπαν ότι δεν μπορούν να χορηγηθούν γρήγορα πολύ τα αρτηματολόγια αυτά για τα απόβλητα. Φυσικά μπορεί να γίνει αυτό σε ψηφιακό επίπεδο. Αναφερθήκαμε και συμπεριλάβαμε και τις συσκευέ αλλιεύσης ε, που δεν συμπεριλαμβανόντουσαν παλιά. Και σε ό,τι αφορά τα τέλη για τα απόβλητα αναλύτρο, τη μεταφορά του στο, στην ξηρά. Ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι αν ε, κάποιος φεύγει από τους ευρωπαϊκούς λιμένες και φεύγει εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης θα πρέπει να παραδώσει όλες του, όλα τα απόβλητα. Εδώ έχουμε κάποιες αμφιβολίες. Μπορεί να είναι μικρός ο λιμένας, μπορεί να μην υπάρχουν σωστές εγκαταστάσεις, να μην υπάρχει δυνατότητα 100% παραδοσής όλων των αποβλήτων. Θα θέλαμε σε κάθε περίπτωση να είναι υπεύθυνο και ο επόμενος λιμένας στο θέμα του κόστους, είναι σημαντικό να τονίσουμε την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Και εδώ είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και την, τον τριμερή διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει 100% ανάθεση, 100% παραδόση. Οι λιμένες είπαν ότι δεν μπορούν δεν μπορεί να είναι αυτό πάντα εφικτό. Εμείς ακολουθήσαμε την οδό του Συμβουλίου. Αυτός ο έμεσος, ε, αυτό το έμεσο τέλος να υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία και το μέγεθος του πλοίου και σε τι αφορά τις μεταφορές ε, και την χωρητικότητα του πλοίου. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Αναφέρεται επίσης και, και τα νερά έρματος ε, ε, να αναφέρονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, συμφωνεί, αλλά εγώ ήθελα να αναφερθεί και στους ορισμούς επίσης είχαμε κάποια ζητήματα. Ως Κοινοβούλιο προτείνουμε κάποιες διευρύνσεις κάποιων όρων. Έχουμε ένα συμβασμό για την τηλογική σκέψη παρελθόν 18. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι ορισμούς εννοούσα στις τελικές σκέψεις διορθώνει η συγγήτρια. Μάλιστα αυτά λίγο πολύ και ελπίζω να μην ξέχασα και τίποτα γιατί προσπάθησα να σας τα πω όλα με χαρτί και καλαμάρι. Αλλά όπως και να έχει να ευχαριστήσω τους κοιόντες συζητητές μου γιατί είναι πάρα πολύ καλή συνεργασία και νομίζω ότι θα πετύχουμε μια φιλόδοξη έκθεση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να ξεκινήσουμε δυναμικά τι διαπραγματεύσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σαφής ε, η παρουσίασή σας, κυρία Μέισνερ. Το λόγο έχει η κυρία Κλούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ για τη δουλειά που έκανε μέχρι στιγμής. Συμφωνώ με τα σχόλια που κάνατε ότι υπήρξε καλή συνεργασία. Τουλάχιστον από το γραφείο μου, με το γραφείο μου και με τους σκιώδεις εισηγητές ε, υπήρξε καλή συνεργασία και αύριο έχουμε άλλη συνεδρίαση των σκιωδών και ελπίζω να υπάρξει πρόοδο. Η κυρία Μάισνερ είπε του τομεί που μα ανησυχούν περισσότερο. Ε, τα πολύ μικρά λιμάνια, τα οποία επιβαρύνονται πολύ από τι διοικητικέ διατυπώσει και έχουν ε, λίγα περιβαλλοντικά ωφέλη. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία με τα μικρά λιμάνια, να μην τα επιβαρύνουμε υπερβολικά με πολλές παραδόσεις, μεγάλες ποσότητες και δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε το κίνητρο το να παραδίνουν τα πλοία, τα απόβλητά τους. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που συζητάμε τώρα. Θα, θα μπούμε σε πολύ έντονες λεπτομέρειες όταν οι ψαράδες παραδίδουν τα παθητικά λιευόμενα απόβλητα δεν θα πρέπει να πληρώνουν γι' αυτό. Θα πρέπει να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στα ενεργά και παθητικά αλλιευόμενα απόβλητα. Επίση, ε, τα πλοία θα, πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν σε τρίτε χώρε, χωρί να πρέπει να παραδίδουν ε, τα αποβλητά του. Ε, θα πρέπει να το δούμε και αυτό το σημείο. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ό,τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και τη γενική νομοθεσία για τα απόβλητα, το, ο στόχος της πρότασης είναι να ευθυγραμμιστεί η ενωσιακή νομοθεσία με τη σύμβαση Μαρπόλ και αυτό κάνουμε. Μ' αρέσει η δουλειά που κάναμε μέχρι στιγμή. Περιμένω τη συνάντηση των σκιωδών αυτή τη βδομάδα και πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόοδο στι λεπτομέρειε. Και ευχαριστώ ακόμα μία φορά την κυρία Μάισνε για τη βοήθεια και την υποστήριξή της. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμμετείχα στην πρώτη συνεδρίαση των Σκιωδών. Θα υπάρξει και νέα συνεδρίαση των Σκιωδών και ευχαριστώ τους συναδέλφους της Επιτροπής ε, Μεταφορών για τη Πραγματικά εργάστηκαν πολύ εργοδός, ε, υπέβαλαν πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ και την ε, γραμματεία. Τώρα, κάποιες σκέψεις. Εν αναμονή των αυριανών διευκρινήσεων. Καταρχάς, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Έχουμε όμως κάποια πράγματα που θα θέλαμε να διαπραγματευτούμε, ούτως ώστε να φτάσουμε σε συμβασμούς. Φέρει πίν. Στην ομάδα μου υπάρχει υποστήριξη για την πρόταση της Κομισιόν για τρία και όχι πέντε έτη. Γιατί είναι μεγάλη η περίοδος η πενταετία μετά από πέντε χρόνια να επαληθεύουμε δηλαδή οτιδήποτε. Γιατί μπορεί να κάνουμε διορθώσεις πολύ νωρίτερα, πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να διαπραγματευτούμε. Ίσως θα μπορούσαμε επίσης να φτάσουμε ε, σε 3 συν 5 δια 2. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποιου όρου. Γιατί, Φερρυπίν, ε, έχουμε υποβάλει τροπολογίε μαζί με τους συναδέλφους για τον ε, όρο της του προγραμματισμένου τρομολογίου ο ορισμός της ε, Κομισιόν δεν μου φαίνεται επαρκής. Εμείς υποβάλαμε ε, τροπολογίες για αυτό τον ορισμό. Υπάρχουν τροπολογίες επίσης για τα οικολογικά πλοία. Είμαστε σύμφωνοι για αυτή την έννοια. Αλλά πώς θα αποφασίζουμε ποιο πλοίο είναι οικολογικό. Γι' αυτό υποβάλαμε τροπολογίες για, αυτή την, ε, για αυτόν τον ορισμό και ελπίζω να γίνουν δεχτές. Επίσης, οι συνάδελφοί μου έχουν υποβάλει τροπολογίε για τον νέο ορισμό των ε, λιμένων. Υπάρχει ένας ορισμός τη Κομισιόν. Εμείς έχουμε μια νέα πρόταση ε, επί κάποιων όρων. Και επίσης, το είπατε κι εσεί. το σύστημα ανάκτησης του κόστους. Θα πρέπει να δούμε το, τη βάση του υπολογισμού, πολύ λεπτομερό. Δεν θέλουμε αυτή η έκθεση να οδηγήσει σε υπερβολικές επιβαρύνσεις για τα μικρά λιμάνια. Θέλουμε να συλλέγονται τα απόβλητα, τα οποία προκύπτουν από τα πλοία, ανεξάρτητα από το είδος του λιμένος. Θέλουμε να μειώσουμε αυτά τα απόβλητα των πλοίων. Άρα θέλουμε μία δίκαιη μεταχείριση και για τη φορολογική επιβάρηση και για τα κίνητρα που δίνουμε, ούτω ώστε να μην ρίχνουμε σημαντικά απόβλητα, βαριά απόβλητα στη θάλασσα. Αυτά είναι κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν όλους τους εισηγητές και τους κοιόδους εισηγητές, γιατί υπάρχουν λιμάνια στις χώρες μας και ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λύση που να είναι εφαρμόσιμη να είναι υλοποιήσιμη. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε πολύ περίπλοκα πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει κανένα. Ευχαριστώ του συναδέλφου για την ε, διαθεσιμότητα να με ακούσουν. Ελπίζω να με ακούσετε και όταν παρουσιάσω με τι τροπολογίε που θα παρουσιάσω εν ονόματι τη ομάδα, ε, γιατί μα ενδιαφέρουν όλου αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο κανονισμό ε, αυτό που έχουμε σήμερα. Ο κύριο Βαντάλεν έχει το λόγο. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε με την επικοδομητική συνεργασία και με την εισηγήτρια και με του κοιόδε. υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινίσουμε για το θέμα τη ε, εσωτερική μα νοσηπλοείας. Η πρόταση αυτή απορρίπτεται Ευτυχώς και χαίρομαι που αναφέρεται και στις ε, απόκεντρες περιοχές η, η συγγήτρια και αναφέρεται στην δυνατότητα ε, επιπρόσθετη εθνική χρηματοδότηση. Είμαστε σε καλό δρόμο, λοιπόν, θεωρώ. Να δούμε το κείμενο τη εισηγητρία όπω το πρότεινε και σε διαφορά κυρίω το άρθρο 2 για την, τον ορισμό και κατά πόσο θα συμπεριληφθεί ο σχετικό ορισμό σε ό,τι αφορά και τα ειζήματα τα οποία προκύπτουν. Για εμένα αυτό αποτελεί σημείο στο οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα εύκολα και να παρουσιάσουμε ποια θα είναι η αποστελικά. Όλες τις Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντάλα Ο κύριο Τέιλ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και Ζήνη. Ευχαριστώ και του υπολείπου σκιώδει για όλε τι παρατηρήσει του για το θέμα αυτό. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα απορρίμματα που βρίσκουμε στις παραλίες και στις, στις ακτές μας και στις θάλασσες μας και που θέτουν σε κίνδυνο το θαλασσιακό σύστημα. Μπορούμε να συζητήσουμε συζητήσαμε ορισμένα από τα κύρια ζητήματα και ορισμένα από αυτά που έμειναν θα τα συζητήσουμε αύριο. Ο βασικός στόχος αυτής της νομοθεσίας είναι να ενθαρρύνει τα πλοία να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των απορριμμάτων στα λιμάνια και γι' αυτό θεωρούμε ότι οποιαδήποτε εξαίρεση ε, δημιουργεί ανησυχία Εάν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα πλοία ε, και όλα τα είδη απορριμμάτων, έτσι ώστε αυτά να φτάνουν στις ακτές, στο λιμάνι και να μην απορρίπτονται στην θάλασσα. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να φτάσουμε σε ένα σύστημα 100% άμεσων ε, τελών, αλλά ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε όχι απλώς ως ένα σύστημα κινήτρων προς τα πλοία. Αντιθέτως, θα πρέπει να αποτρέπουμε με αποτελεσματικό τρόπο την απόρριψη των απορριμμάτων στη θάλασσα. Θα πρέπει κατά την άποψή μας λοιπόν να ποινικοποιηθεί η απόρριψη των ε, λιμάτων αυτών στη θάλασσα. Γιατί είναι κρίσιμη σημασία για να έχουμε ε, καθαρές θάλασσες. Γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στα απορρίμματα που, που ρίχνονται, στη θάλασσα είναι και ε, εργαλεία αλλιευτικά, τα οποία καλύπτονται ήδη από κανονισμό του 2009. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, με έκπληξη, έκπληξη πίστοσα ότι διαγράφεται αυτή η υποχρέωση που είχαν οι, τα πλοία να ε, επανακτούν τον, τα αλλιευτικά εργαλεία που είχαν χάσει μέσα στις 24 ώρες. Καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις που είχαν και συνεχίζουν να έχουν μέχρι τώρα να ενημερώνουν και να ε, περακολουθείτε αυτό το φαινόμενο σε ολόκληρο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα πίσω γύρισμα το οποίο έχει ανησυχήσει την κοινωνία των πολιτών, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε αποτελεσματικά στοιχεία, ουσιαστικά στοιχεία μάλλον, για τα αλλιευτικά εργαλεία που απορρίπτονται στην θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο το λόγο λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους συναδέλφους το θέμα αυτό των αλληλευτικών εργαλείων να καλυφθεί. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και αύριο. Ευχαριστώ κύριε Κονζάλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνε για την απόλυτη και αμέριστη βοήθεια για τις εργασίες εργασίες. Ε, να συνοψίσω τις τροπολογίες οι τυχαίες επιθεωρήσεις, οι κυρώσεις θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται όπως και τα εγκλήματα κατά της δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει να ρίχνουμε επίσης λίματα ή λίματα ε, έρματος ή από πλυντρίδες ε, στην θάλασσα. Επίσης, η λιματα ερματος η απο πλυντριδες στην θαλασσα επισης υποχρέωση στον καπετάνιο του αλληλευτικού σκάφου, σε περίπτωση που χάνουν αλληλευτικά εργαλεία, να ενημερώνει πολύ σύντομα. Να έχουμε κανόνες ε, για τα αλληλευτικά σκάφη. Επίσης, η κατάρτιση και η ενημέρωση των εργαζομένων ε, και των λιμενικών σε σχέση με τα καθήκοντα της αποκατάστασης, καθαριότητας, η διαχείριση των ε, της μεταφοράς ε, επιβατών και φορτίων ε, και να δημιουργήσουν εθνικά ταμεία για υποστήριξη όλων αυτών των δράσεων. Επίσης, υπάρχει συμβιβασμό της Κομισιόν για τα περιβαλλοντικά θέματα, για τον καθορισμό ε, ενό ορισμού Μιλάμε για τη συμβαστική παριθμόν 7, η οποία μιλάει για τον ορισμό των αποβλήτων σκαφών. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος βάζει τον ορισμό πλατφορμών ε, σταθερών ε, ή που επιπλέουν με την υποστήριξη των πρασίνων. Είναι σημαντικό να βάλουμε αυτόν τον ορισμό στην εκθεσή μας και τέλος, κάτι που είχαμε σχολιάσει σε κάποιες περιπτώσεις, το μέγεθος των λιμένων που εξαιρούνται. Ο ορισμός των μικρών και πολύ μικρών λιμένων, ποιοι είναι, να δούμε ποιο είναι το μέγιστο, μέγεθος που πρέπει να έχει ένα πλοίο, ώστε να έχει ένα σχέδιο ε, παραλαβής και να είναι ανεξάρτητο αυτό από τις, α, από τις τοπικές αρχές. Ε, εμείς στο Μπιλμπάο για τα μικρά λιμάνια μπορούμε, ε, έχουμε προβλέψει μάλλον να συνεργάζονται τα μικρά λιμάνια, αρχές των μικρών λιμένων, τόσο ώστε να έχουν κοινά σχέδια για την παραλαβή. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά συνενετικά σημεία στην έκθεση και ελπίζουμε οι τροπολογίε μα να ενσωματωθούν ε, στην έκθεση ή σε συμβαστικέ τροπολογίε. Ευχαριστούμε πάντω την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. Ε, ευχαριστούμε του υπόλοιπου σκιώδει εισηγητέ για την καλή του διάθεση να συνεργαστούν. Και ελπίζω αύριο το πρωί να μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποια κενά που ακόμα εκκρεμούν. Ευχαριστώ. Και τώρα η Κομισιόν έχει το λόγο. Η κυρία Μπέργκ. Και σας καλωσορίζω και στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ και όλους τους σκιώδης ηγητές για τη δουλειά που κάνανε για το θέμα αυτό, που τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα απόβλητα από τα πλοία φτάνουν στα λιμάνια και δεν απορρίπτονται στη θάλασσα. Και τα αποβλήματα, τα απόβλητα ε, τα οποία ψαρεύουν τα ληφτικά δίχτυα και αυτά να καταλήγουν στα λιμένια χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον οι ψαράδες. Επίσης, θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για την επίσκεψη της κυρίας Μάισνερ στην ΕΝΣΑ και η πρόεδρος θα ήθελε να είναι εκεί. Σας χαιρετίζει πάντως ο κύριος Μίλη. Όπως εξηγούς, πάντα έχουμε πει, η πρόταση της Κομισιόν έχει εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με την ΕΜΣΑ, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο ε, στην εφαρμογή της ε, πρότασης που θα προκύψει, της νέας πρότασης. Να εστιάσω σε τρία θέματα, τα οποία είναι τα πιο σημαντικά και αντικατοπτρίζονται και στις τροπολογίες, καθώς και στις συμβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν. Αυτό αφορά καταρχάς το έμεσο τέλος 100% ε, για τα σκουπίδια και τον περιορισμό του όγκου των αποβλήτων, ε, το θέμα των παθητικά αλλιευόμενων ε, αποβλήτων, που είναι ένα όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στα θάλασσές μας, και τέλος την κατάσταση των μικρών και πολύ μικρών λιμανιών και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μάισνερ. Είναι μια οδηγία αυτή που προσπαθεί να εξασφαλίσει την εναρμόνιση, αλλά είναι δύσκολο να καλύψουμε τα πάντα. Αν είμαστε σοβαροί για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων αποβλήτων από τα πλοία, θα πρέπει να έχουμε και σωστά οικονομικά κίνητρα, ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή παραλαβή των αποβλήτων από τα πλοία στην ακτή. Και τα ε, τέλη που με βάση τον όγκο, κατά τη γνώμη μας, και με την αξιολόγηση που κάναμε, δείχνει ως αντικίνητρο για την παράδοση. Γι' αυτό, με αυτό το 100% έμεσο φόρος, ε, τέλος για τα απόβλητα, πιστεύουμε ότι δημιουργούμε το σωστό αυτοκίνητρο, αλλά θα θέλαμε ότι και τα λιμάνια θα μπορούν να διαφοροποιούν το τέλος αποβλήτων με βάση το μέγεθος του πλοίου, τη χωρητικότητα και τα μοντέλα εμπορίου. Δεν είναι μία 100% εναρμόνιση σε όλη την Ευρώπη μέσω αυτής της οδηγίας που επιδιώκουμε. Επίσης, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο δίδουμε αρκετά κίνητρα στα λιμάνια για να επενδύσουν σε επιπλέον υποδομές, ούτω ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων και να μπορούν αυτά να παραδίδουν τα αποβλητά τους στα λιμάνια που επισκέπτονται. Για τον περιορισμό του όγκου των αποβλήτων που συζητήθηκε μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά πιστεύουμε και ελπίζουμε αυτός ο περιορισμός του όγκους να γίνεται μόνο σε περίπτωση κάποιων εξαιρέσεων. Εκεί δηλαδή όπου τα πλοία, τα οποία θέλουν να παραδώσουν περισσότερα απόβλητα από όσα δηλώνουν στο, δυναμικό χωρητικότητά τους, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα πληρώνουν επιπλέον ούτως ώστε ο περιορισμός του όγκου να μην καθορίζεται από τα λιμάνια. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις στα λιμάνια. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε το σημερινό μοντέλο που δημιουργεί πάρα πολλέ διαφορετικέ πραγματικότητες από λιμάνι σε λιμάνι και δεν δίνει και κανένα κίνητρο στα λιμάνια για να επενδύσουν σε νέε υποδομέ. Γιατί θα πούνε πολύ γρήγορα, «Α, αυτό είναι εξαιρετικό, είναι επιπλέον ποσότητα, παραπάνω ποσότητα από αυτή που θα παραδίδεται, άρα πληρώνεται για αυτή. Ελπίζουμε λοιπόν να βρεθεί ένα καλό συμβασμό για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τα παθητικά αλλιευόμενα απόβλητα, αυτά που καταλήγουν δηλαδή στα λιευτικά δίκτυα, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η πρότασή μας δίνει στους ψαράδες το δικαίωμα της παράδοσης ε, εφόσον πληρώσουν ένα τέλος, το οποίο ούτως ή άλλως το πληρώνουν και σήμερα. Και επιπλέον, ε, και τα κράτη-μέλη κρατούν την ελευθερία τους για να χρησιμοποιούν τα έσοδα από άλλα προγράμματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή, όπως ε, η παρατεταμένη ευθύνη των παραγωγών, ας πούμε, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οποιοδήποτε επιπλέον κόστος το οποίο προκύπτει για τα λιμάνια θα αντισταθμιστεί ε, από τα έσοδα από αυτά τα τέλη. Το θέμα των πολύ μικρών και μικρών μη εμπορικών λιμένων, το τελευταίο θέμα. Και ανησυχούμε για μια γενική εξαίρεση για όλα τα μικρά λιμάνια να μην ε, έχουν καθόλου δηλαδή, ένα σχέδιο για τα ε, ένα σχέδιο για τα απόβλητα και να, που να, πρέπει να το κοινοποιούν στο κοινό και να ενσωματώνουν αυτό το σχέδιο για τα απόβλητα στις ε, δημοτικές ε, υποδομές. Αυτή η εξαίρεση μας ανησυχεί, επαναλαμβάνω. Το να είσαι μικρό λιμάνι δεν σημαίνει ότι δεν δίδεις κάποιες δεν κάνεις κάποιες υπηρεσίες. Και εφόσον ε, κάνεις κάποιες υπηρεσίες και παίρνεις λεφτά, ας πούμε, θα πρέπει να δίνεις και ένα τιμολόγιο για αυτό που χρεώνεις. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους βουλευτές, ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η πρόταση. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ja, ich glaube, ich kann das relativ... Ε, κυρία Μάιστερ, θα είμαι σύντομη και άκουσα με μεγάλη προσοχή και κράτησα σημειώσει. Τα λέμε αύριο το πρωί. Έχουμε δύο ώρε ε, για να διευκρινίσουμε τα εκκρεμή ζητήματα και να δούμε ποια θα είναι η οριστική μα τοποθέτηση. Το θέμα των τριτών κρατών Ευρωπα... εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ενδεχομένω να το δεχτούμε. Για το green shipping, ναι, έχουμε βρει ορισμό και κάποια στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμβιβασμό, αλλά νομίζω ότι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, διευκρινίσαμε κάποια πράγματα και το θέμα των αποβλήτων. Θα πρέπει να ξέρουμε στους ορισμού ε, τι γίνεται για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Πώς θα υπάρξει ενιαία διαμόρφωση στα κράτη-μέλη. Φυσικά και εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπάρχουν άλλα απόβλητα στι θάλασσε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι ισχύει για τι εξαιρέσει. Όλα θα πρέπει να μεταφέρονται στη ξηρά λοιπόν και σε ό,τι αφορά τους μικρού λιμένε θα πρέπει να δούμε πώ θα τα καταφέρουμε. Σε ό,τι αφορά τι πετρελαϊκέ πλατφόρμες τώρα. Ξέρω. Και το συζήτησα και με τον Μπασάικοτ. Συμμετείχε και σε διάφορες συνεδριάσεις των σκιωδών. Φαίνεται ότι δεν ε, λειτουργεί, γιατί ε, μεταφέρουν τα πλοία οι πλατφόρμες αυτές, αλλά όχι απόβλητα. Δεν μπορούν να μεταφέρουν ε, τα απόβλητα στην ξηρά, αφού το κάνουν τα πλοία. Άρα δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Το συζητάμε όμω και αύριο. Για τις εξαιρέσει θα πρέπει να παραμείνουν σε ελάχιστο επίπεδο και θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι και στους μικρούς λιμένες που θα ε, Ξερούνται ενδεχομένω να υπάρχει συνεργασία και να συμπεριλαμβάνεται και το τοπικό σύστημα λιμάτων ή ε, ή εν πάση περιπτώσει να το αποδείξει αυτό, να το αποδεικνύει αυτό το κράτος μέλος και σε ό,τι αφορά του περιορισμού, σε ό,τι αφορά το τέλος 100% ε, φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ συναρπαστικά στους τρεμερούς διαλόγους, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Το βασικό βέβαια είναι ότι όλοι συμφωνούμε να μεταφέρουμε τα αποβλητά στην ξηρά. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Ευχαριστώ πολύ εκεί Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 28 ε, Οκτωβρίου. Στις 29 Οκτωβρίου. Τώρα, μια απόφαση για το Ταμείο Συνοχής και για το θέμα των, ε, της δημιουργίας κανόνων για το ταμείο αυτό σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια για ένα άμα τέτοιο ταμείο για το αγμείο ασύλου και μετανάστευση, ταμείο ιστορικής ασφάλειας και το μέσο για τη χρήση των συνόρων Ο εισηγητής μας είναι ο κ. Λουτόφσκι και έχει το λόγο. Merci, Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι από τον τίτλο και μόνο αυτού του κανονισμού, πόσο μεγάλη είναι η σημασία του, είναι τόσο μεγάλο ο τίτλο που είναι δύσκολο να τον θυμάται κανεί. Αλλά είναι ένα, θέμα, είναι πολλά θέματα μάλλον τα οποία σχετίζονται με την πολιτική συνοχή και με την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, η συζήτηση για το πολιτέ νομικό πλαίσιο θα επηρεάσει και αυτό το τομέα και αυτού του τομεί. Στόχο του κανονισμού αυτού είναι να μειωθεί το άχθος, το διοικητικό και έτσι να είναι πιο αποτελεσματική η χρήση των δημοσίων πόρων. Είναι ένα στόχος αυτός που όλοι υποστηρίζουμε. Ωστόσο, ήδη κανείς μπορεί να αναφέρει, ότι δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί να πρέπει να μειωθεί στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο η χρηματοδότηση για τις περιφέρειες μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό ερίστον παρόλο. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2020-2027 θα πρέπει να ε, παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με το τρέχον, τουλάχιστον όσον αφορά τις υποδομές. Ε, αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβω εδώ όλα τα επιχειρήματα γιατί είναι σημαντικό. Θα αναφερθώ όμως σε κάποιες αλλαγές που κατά την άποψή μου είναι απαραίτητες, αλλαγές δηλαδή στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, η διαφοροποίηση που έχουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ των πόρων ε, που θα μεταφερθούν από τα ταμεία ε, υποδομής προς, τα, προς το Ταμείο Connecting Europe. την άποψή μας, αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε εθνικούς, ε, στα, στα κράτη-μέλη και μετά να γίνονται προκηρύξεις για τα διάφορα έργα. Επίσης θέλουμε να διατηρηθεί η χρηματοδότηση από το 80% από το 70% για τις περιοχές της λιγότερο αναπτυγμένες. Γιατί ήδη έχουν αναλυφθεί υποχρεώσεις σε αυτές τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και μια τέτοια μείωση μπορεί να οδηγήσει σε, ε, στο να σταματήσουν ορισμένα project. Και αυτό θα είναι απαράδεκτο γιατί θα σταματήσουν οι επενδύσει ακριβώ εκείνε τι περιοχέ που είναι πλέον απαραίτητε και ακριβώ εκείνε τι επενδύσει που είναι πιο δύσκολο ε, να βρεθεί χρηματοδότηση για αυτέ. Αυτή τη στιγμή έχουμε το σύστημα N3, το οποίο λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά, έχει αποδείξει την αξία του και σε πολύ ε, περίπλοκα ε, έργα τα οποία χρειάζονται τη σχεδιασμό πρόταση της Επιτροπή να περάσουμε σε ένα σύστημα ενίσυν 2, στην πραγματικότητα απλώ θα περιπλέξει τα πράγματα για τα κράτη-μέλη και για τις περιφέρειες, χωρίς στην πραγματικότητα να βελτιώσει τη χρήση των δημόσιων πόρων. Το μόνο που θα δημιουργήσει θα είναι ε, απώλεια πόρων. Τώρα, όσον αφορά τη σύνδεση ε, της, χρηματοδότησης με τον σεβασμό του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος. Αυτό μας ανησυχεί, μας ανησυχεί να μην χρησιμοποιείται με τρόπο που να το καθιστά ένα πολιτικό εργαλείο και δηλαδή με έναν τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με τη χρηστή διοίκηση ή τη χρήση των πόρων. Αυτό το θέμα εμεί το θεωρούμε πολύ σημαντικό, μιας και μιλούμε για μια πολιτική μακρόπνοη. Αυτά από την πλευρά μου. Περιμένω τις τροπολογίες σας, τις προτάσεις σας έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια ουσιαστική ε, πρόταση προς την Αρμόδια Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε Ζλωτόφσκι για την παρουσίαση της εκθεσής σας. Ο κύριος Φαντερκάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, της ομάδας ε, του ΕΛΚ είμαι ο σταθερός εκπρόσωπος στη σημερινή συνεδρίαση και έχω την τιμή να εκπροσωπώ την ε, συναδελφό μου την κυρία Κλάουντια Σμίτ από την Αυστρία για το θέμα αυτό. Η κυρία Σμίτ θέλει να βγουν αυτά από τις χώρες συνοχής ε, και έχουμε υπόψη να ε, Μάλλον έχουμε λίγο μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτική συνοχή σε σχέση με τον κύριο Σλοντόφσκι, ο οποίο λίγο πολύ θέλει να μείνουν τα πράγματα όπω ήταν στο παρελθόν και θέλει να αυξηθούν τα κονδύλια για τα ταμεία συνοχή. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση θα είναι πολύ δύσκολη. Γιατί λάβαμε και μια πολύ επικριτική έκθεση του ελεκτικού συναντρίου σε ό,τι αφορά την ανάθεση κονδυλίων από τα μία συνοχή στα περιφερειακά αεροδρόμια σε υπερταχείες συνδρομικές γραμμές και την εφαρμογή του ERTMS. Το ΕΛΚ ε, πρέπει να ξέρετε ότι δίνει μεγάλη αξία στα ταμεία συνοχής και στα σχετικά κονδύλια και σε ό,τι αφορά λοιπόν και αυτές τις ε, γενικές διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες θεωρούμε ότι μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη επικριτική διάθεση για το πώς πάνε τα κονδύλια από τα Ταμεία Συνοχής. Το ότι συγκαταλέγονται απλά στις εθνικούς φακέλους είναι... δεν είναι αρκετό, πιστεύουμε. Η ομάδα μας λοιπόν συζητά την πρόταση 30%-70% υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, υπάρχουν και διάφοροι πιο επικριτικοί συνάδελφοι σε ό,τι αφορά τη διατύπωση των όρων για την ανάθεση των κονδυλίων. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι διατείνονται ότι κοιτάξτε, εφόσον πρόκειται για ταμεία συνοχή, θέλουμε να τα βάλουμε στι μεταφορέ, πρέπει να μα αφήσετε να κάνουμε αυτό που θεωρούμε το πιο κατάλληλο. Εν συντομία, ο κανονισμό αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δαπάνη όμως των κονδυλίων ε, συνοχής μπορεί να είναι λίγο πιο μαζεμένη. Γιατί τα χρήματα αυτά μία φορά θα τα δαπανίσουμε. Θέλουμε φυσικά μεγαλύτερη επικέντρωση στο δίκτυο TNT, αλλά και εγώ και η κυρία Κλάουντια Σμιτ θεωρούμε ότι συνολικά η προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα φάση δεν είναι η ενδεδειγμένη. Ευχαριστώ. pour le... Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Κύριε Σιγητά, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν, θα υπάρξει ομόφωνη στήριξη, φαντάζομαι, για τις προτάσεις που έχουν σαν στόχο να μειώσουν την γραφειοκρατία και το περιττό, τις περιττές σπατάλες ε, των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Επίσης, θα πρέπει να είναι πιο εναρμονισμένοι οι κανόνες των διαφορών ταμείων, ούτως ώστε τα ταμεία να παίζουν συμπληρωματικό χαρακτήρα για να υλοποιεί το ίδιο στόχος. Αυτά είναι θετικά στοιχεία και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε στην Κομισιόν ότι δεν θα βάλουμε εμπόδια, δεν θα βάλουμε φραγμού σε αυτά. Σε ό,τι αφορά τη σύγκληση μεταξύ κρατών και περιφερειών, σε διάφορα σημεία του κειμένου αναφέρεται αυτός ο στόχος. Είναι κρίμα όμως που αυτές οι ενδείξεις δεν συνοδεύονται από το απαραίτητα κονδύλια. Είναι περίεργο που μας παρουσιάζει η Κομισιόν ένα κείμενο το οποίο εκφράζει την ανησυχία της και την διάθεσή της ανάμεσα ε, για την έλλειψη ε, σύγκλησης ανάμεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά κόβει κατά 45% τα κονδύλια για αυτό το στόχο. Ε, μην ξεχνάτε πόσο αρνητικά μας βλέπουν οι πολίτες ε, σε σχέση με αυτό το θέμα, το, τον τρόπο χρήσης των κονδυλίων, των ταμείων δηλαδή. Εγώ είμαι Πορτογάλος. Και συχνά οι επενδύσεις που έχουν κάνει η πολιτική μας ε, έγιναν για να ανακτήσουμε την καθυστέρηση που είχαμε για διάφορους λόγους. Η Ευρώπη μας βοήθησε, βοήθησε το κράτος Πορτογαλίας. Το αναγνωρίζει αυτό η χώρα μας και πολλοί κάτοικοι ε, είναι υπέρ της Ευρώπης και υπέρ των ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων. Είναι ανησυχητικό όμως που η Κομισιόν προβλέπει μείωση της ευρωπαϊκής ε, συγχρηματοδότησης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα υπάρξει μία μείωση ε, στην εκτέλεση των προγραμμάτων ε, και στον τομέα των μεταφορών, που είναι όμως πολύ σημαντικά για να προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτών των περιφερειών, των λιγοτών επιτυγμένων δηλαδή. Δεν συμφωνώ με την σύνδεση ανάμεσα στον ε, αποκλεισμό των ευρωπαϊκών ταμείων και σε σχέση με το κράτος δικαίου, δηλαδή για λόγους εφαρμογής των αρχών κράτους δικαίου. Ε, Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία κατ' επανάληψη ε, παραβιάζουν ε, το κράτος δικαίου. Και παρόλα αυτά συνεχίζουν να παίρνουν κονδύλια. Είναι πολύ σημαντικές οι αρχέ του κράτους δικαίου, ίσως πιο σημαντικές από, την, από τον σεβασμό των, των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα που πλήττουν την Ευρώπη εδώ και 10 χρόνια ουσιαστικά. Και μερικές φορές, παρότι κάποιες κυβερνήσεις είχαν τη θέληση, δεν ε, μπόρεσαν να σεβαστούν τους στόχους για την εξορρόπηση ε, των δημοσιονομικών και για αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, αυτό όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Θα υποβάλουμε τροπολογίε για να βελτιώσουμε την πρόταση που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Από το Άλντε θα πάρω εγώ το λόγο. Αυτό που ήταν ένας μηχανισμός ε, για την ε, κατανομή των ε, κονδυλίων των ταμείων μπαίνει σε μία δυναμική που τελικά συν το χρόνο επηρέασε τα διάφορα κράτη-μέλη. Και λόγω της οικονομικής κρίσης που την ανέφερε ο κύριος Ασής, αλλά και λόγω της πολιτικής κρίσης που επίσης αναφέρθηκε. Επομένως, υπάρχουν κάποιες ποσοτικές και κάποιες ποιοτικές αλλαγές ε, που γίνονται. Η συζήτηση ε, γίνεται σε εθνική βάση. περισσότερο σε εθνική βάση παρά σε πολιτική βάση από ό,τι βλέπουμε εγώ. Καταρχάς, ό,τι αφορά την έκθεση Ισλοτόφσκι, συμφωνώ με κάποιες από τις παρατηρήσεις του. Καταρχάς, φυσικά θα δούμε... Θα συμφωνούμε με την Κομισιόν ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, μείωση του γραφειοκρατικού άχθους, ε, ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων, ε, κάποια πράγματα τα οποία δηλαδή πηγαίνουν προς την καλύτερη διαχείριση και τη μεγαλύτερη συνέπεια ε, με βάση τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ε, παραμένει ένα μόνιμο πρόβλημα, μια διαφορά ανάμεσα στις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα αιτήματα των κρατών μελών, ειδικά τα κράτη-μέλη της συνοχής, για τη δική τους διαρθωτική ανάπτυξη ή την ανάγκη να καλύψουν κάποια διαρθωτική υστέρηση που έχουν. Το πρώτο πρόβλημα, και εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή, εγώ θα κρατήσω το μηχανισμό κατανομής των κονδυλίων των ταμείων συνοχής. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, μεγάλη σύνεση. Η μείωση των κονδυλίων, του όγκου. Αυτό θα πρέπει να το δούμε με βάση την, πολιτική της, με βάση την κατεύθυνση της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή η διαρθρωτική ανάκτηση του χαμένου χρόνου των κρατών ε, θα πρέπει να δούμε και τι προσπάθειες κάνουν οι χώρες συνοχής, τι αποτέλεσμα έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, ε, αλλά αν τα συμβολογήσουμε όλα αυτά, αυτή η καθυστέρηση έχει μειωθεί. Τα ειδικά μέτρα για να ανακτηθεί ο, ο χαμένος χρόνος πρέπει να ειδωθεί σε σχέση με τα νούμερα. Αυτή η καθυστέρηση μειώνεται όμως. Ε, όταν μειώνεται η καθυστέρηση θα πρέπει να μειώνεται και τα κονδύλια των ε, ταμείων. Δηλαδή, αν αυξήσουν τα... Αν αυξάνονταν τα κονδύλια των ε, ταμείων ή παρέμεναν σταθερά, θα ήταν ε, απελπισία η κατάσταση. Σημαίνει ότι δεν ανακτούν το χαμένο χρόνο τα κράτη συνοχή. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Θα μειώνουν τα κρατη συνοχης επομενως θα πρεπει όσο αυξάνεται ε, η ευθυγράμμισή τους με τα υπόλοιπα χρόνια. Επίσης, ε, το μέτρο για την εκμετάλλευση. Είμαστε στα πλαίσια του refit. Αυτό είναι ένα μέτρο που αύξησε την περιπλοκότητα και το διοικητικό άχθος ε, για τους φακέλους. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο δικαιολογείται θεωρητικά αλλά κατά πάσα πιθανότητα ε, θα το μισήσουν όσοι ασχολούνται στην πράξη με αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην αρετή και, την, ε, και το ρεαλισμό, και την, πρακτική πτυχή. Συμφωνώ με τον εισηγητή για αυτό το θέμα και ε, συμφωνώ με την αποψή του για τα ποσοστά και τα αρχικά ποσά. Αν οι χώρες συνοχής θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα και πρέπει να δούμε τα πολύ μικρά αρχικά ποσά. Ο εξορθολογισμός του προγραμματισμού. Αυτό θα μειώσει ε, το φόρτο. Είναι καλή ιδέα. Αντίθετα από την ιδέα που είχαν οι προηγούμενες μελέτες για τις δαπάνες και τα λοιπά, θα, νομίζω θα είναι ένα θετικό πράγμα. Πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, δύο οικονομικές παρατηρήσεις. Πρέπει να το βάλουμε αυτό στο γενικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Το βασικό είναι το πουδουπού. Θα πρέπει να γίνουν πολλές... Θα υπάρξουν διάφορα, διάφορες δούνε και λαβίνα. ας πούμε, ε, διάφορα, θα υπάρξει μια διαιτησία ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις. Επανέρχομαι στο, στα 20 δις, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με αυτό που θέτουν οι σχετικοί κανονισμοί και οι οδηγίες. Ο κ. Τέιλορ από τους πράσινους δεν θέλει να πει τίποτα. Όχι, από ό,τι βλέπω. Άρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζηλό από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιου που θα εκπροσωπήσει την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την... και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για το προσχέδιο έκθεσης και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου για τη σημερινή συζήτηση. Ναι, θα αναγνωρίσω κι εγώ ότι ο τίτλος της έκθεσης του κανονισμού είναι μακροσκελής. Όμως, θα πρέπει να τονίσω ότι ο προτινόμενο κανονισμός είναι κατά 50% ε, μικρότερος, βραχύτερος από τον υφιστάμενο. Τώρα, το να κόψει κανείς το, το, κανονισμό, το κείμενο του κανονισμού στο μισό δεν σημαίνει ότι έχουμε αμέσως απλοποίηση. Ωστόσο, ε, πολλά μέλη της Επιτροπής σας αναγνώρισαν ότι πράγματι υπάρχει μια ε, απλοποίηση, μεγαλύτερη ευελιξία και αυτό επιδιώξαμε να το ε, καταφέρουμε με όλα τα στοιχεία της πρότασής μας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα από τις ε, παρατηρήσεις που είναι. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει μια κάποια αντίφαση. Γιατί αφενός λέμε ότι μας ανησυχεί που ο προπολογισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα για τα ταμεία συνοχής, είναι χαμηλότερος και αφετέρου να ζητείτε να αυξηθεί ο συντελεστής συγχρηματοδότησης. Γιατί αυτό που εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε ως ιδέα είναι ότι αν υπάρχει χαμηλότερη συγχρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό οδηγεί ώστε το, το έργο να είναι μεγαλύτερο ενδιαφέροντος και να ε, ε, επενδύει σε αυτό περισσότερο το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε αυτή την θετική εμπειρία που ακούστηκε ότι υπήρχε με το σύστημα N3 κατά την άποψή μας αυτό ήταν ένα από, τις, ε, από τους σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν σε καθυστερήσεις κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Και ήταν και μία από τις προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όταν προσπαθήσαμε να υπολογίζουμε για την επόμενη προγραμματική ε, περίοδο της προχρηματοδοτήσης. Γιατί τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα από τα τρέχοντα προγράμματα κατά την περίοδο 2020-2023 είναι τόσο πολλά, είναι τόσο υψηλός αυτός ο βαθμός που μας ε, έδαινε τα χέρια για την χρηματοδότηση προγραμμάτων έως το 2027. Με άλλα λόγια, οι καθυστερήσεις που διαπιστώνουμε τώρα θα ε, γνωρίζουμε ήδη από τώρα ότι θα έχουν ε, θα δημιουργήσουν προβλήματα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να σταματήσουμε το σύστημα νησιν 3 και να πάμε σε ένα σύστημα νησιν 2. Μετά, ακούστηκε ότι η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει την απέτηση να καλύπτονται τα έξοδα ε, συντήρησης και λειτουργίας υποδομών. Θα ήθελα να σας εξηγήσω τι γίνεται εδώ. Εδώ προσπαθούμε να έχουμε ένα στρατηγικό ε, να δημιουργείται μάλλον ένα στρατηγικό σχέδιο στην αρχή της προγραμματικής περίοδου, το οποίο να αποδεικνύει ότι το κράτος μέλος έλαβε υπόψη του τα έξοδα ε, συντήρησης και λειτουργίας για τις υποδομές τις οποίες προτείνει να χτίσει, προτείνει να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια τη ε, προγραμματική περίοδου. Αυτό δηλαδή δεν είναι ένα τρόπο για να δημιουργήσουμε καθυστερήσει ή να επιβάλλουμε κάτι, αλλά προσπαθούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να μας εξασφαλίσουν ότι δεν θα ασχοληθούν μόνο με το αρχικό κόστος της δημιουργίας μιας υποδομής, αλλά θα έχουν να ασχοληθεί επίσης και με το πόσο εθνικός τους προπολογισμός από εκεί και πέρα θα καλύψει τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης του έργου. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σλοτόφσκι, τον εισηγητή μας. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω σε αυτή την έκθεση. Θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται περισσότερο εξορθολογισμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση αυτών των πόρων. Των πόρων από αυτά τα ταμεία. Νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι. Ο σκιώδη συζητητή από την Πορτογαλία, κ. Σασή, μα έλεγε ότι ίσως να υπάρχουν κάποιες χώρες, κάποια κράτη-μέλη τα οποία να μην σέβονται το κράτος δικαίου και αυτό να έχει επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση, στην ε, υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων. Πρώτα απ' όλα, κύριε συνάδελφε, τι σημαίνει ακριβώ μια χώρα να σέβεται το κράτο δικαίου. Κατά την άποψή μου εδώ θα χρειαστεί να υιοθετήσουμε έναν ορισμό αυτή τη έννοια, τουλάχιστον για του σκοπού τη έκθεση. Δεύτερον, υπάρχουν κάποια προγράμματα, κάποια έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία τα ευρωπαϊκά για τα οποία συζητούμε. Σε αυτέ τις περιπτώσει Ε, δεν έχει υπάρξει καμία σκιά όσον αφορά την ίδια την επένδυση. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο μου φαίνεται τρελό να συζητούμε για σεβασμό του κράτους δικαίου. Όταν έχουμε ένα περιφερειακό αεροδρόμιο και χτίζουμε 20 χιλιόμετρα από αυτό ένα άλλο περιφερειακό αεροδρόμιο, αυτό από οικονομικής απόψεις είναι ηλίθιο και δεν έχει καμία σχέση με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα περιφερειακό αεροδρόμιο κοντά στο Γκτάνσκ και χτίστηκε ένα νέο περιφερειακό αεροδρόμιο 20 χιλιόμετρα από αυτό. Από την πλευρά του κράτους δικαίου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά κατά την άποψή μου αυτό που έχει παραβιαστεί εδώ είναι η κοινή λογική. πού πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, εστιάζει αυτός ο κανονισμός, ποιο θα πρέπει να είναι η πιο σημαντική του επιδίωξη. Να γίνονται επενδύσεις οι οποίες στην ουσία να βοηθούν στην συνοχή, να συνεισφέρουν στην βελτίωση της συνοχής και να μην γίνονται σπατάλες. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το εάν μια χώρα ε, σέβεται ή δεν σέβεται το κράτος δικαίου συνέβησαν περιστατικά να έχουν χρηματοδοτηθεί έργα με το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα οποία ήταν παράλογο να χρηματοδοτηθούν και αυτό ελπίζω να μην επαναλήφθει. Προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε, προσβλέπω στις τροπολογίες έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Θα σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Συγγνώμη διορθώνει η πρόεδρο. dépôt est fixé le 5 octobre. 5 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Σα τρόμαξα λίγο. Και 15 Νοεμβρίου στην Επιτροπή η ψηφοφορία. Το λόγο όμω έχει ο κύριο Σωσή. Θέλετε να πάρετε το λόγο και πάλι. Ναι, θα ήθελα να διευκρινίσω μόνο το εξή, αν με επιτρέπετε. Ξέρω τι είναι το κράτος δικαίου, ξέρω και πώς ορίζεται το κράτος δικαίου. Αυτό ορίζεται και στις ευρωπαϊκές συνθήκες, Άλλωστε, δεν είναι σωστή στιγμή ωστόσο να το συζητήσουμε αυτό. Και πάνω απ' όλα, ξέρω ακριβώς τι σημαίνει να μην ακολουθούνται οι κανόνες του κράτους δικαίου. Γιατί δυστυχώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε κάποιο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αυτοκρατικά καθεστώτα με δημογραφικό πρόβλημα και αυτό είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι οι χώρες αυτές που δεν ακολουθούν το κράτος δικαίου θα πρέπει να γνωρίσουν και οικονομικές κυρώσεις. Όχι απλά επειδή μπλέκουμε δηλαδή το θέμα του κράτου δικαίου με τα οικονομικά προβλήματα. Ένα δεύτερο ζήτημα. Φυσικά θα πρέπει να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε το πώς έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν μέσω των ε, μηχανισμών ε, ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμοστούν 100%. Ε, και ήθελα απλά να διευκρινίσω τι εννοούσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Λοτόφσκι, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε συζήτηση ε, για το κράτος δικαίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που γνωρίζει ο συνάδελφο τι είναι κράτος δικαίου. Και εγώ το γνωρίζω. Υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν ακολουθούν το κράτο δικαίου, είπατε. Θέλετε όμω να τι απαριθμίσετε. Και ποια είναι η παραβίαση του κράτου δικαίου, το οποίο, την οποία εσείς έχετε να καταγγείλετε. Κλείνεται συζήτηση, λέει η Πρόεδρος. Αν θέλετε να κάθετε να συζητήσετε τα περί κράτου δικαίου, πάτε να πιείτε ένα καφέ. Δεν αποτελεί αυτό το αντικείμενο της έκθεσης. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι η πρόταση για την κατάσταση τροπολογίων είναι η 5η Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι για να ψηφίσουμε 15 Νοεμβρίου και συνεχίζουμε για ένα, με ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά την έκθεση εφαρμογή, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό 1-2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο εισηγητής μας για το σχέδιο προς την Επιτροπή Πολιτισμού είναι κύριος ε, Keith Taylor, ο οποίος και έχει το λόγο. Uh, well, thanks, Jim. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίζω αυτή την ευκαιρία ως εισηγητής ε, να συζητήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής Μεταφορών το θέμα αυτό της έκθεσης εφαρμογής και είναι η αρμοδιότητα μεταξύ ενβί και ΤΡΑΝ και ΑΓΡΙ σε ό,τι αφορά τις διάφορες πτυχές των αρμοδιοτήτων των εκάστοτε επιτροπών. Σε ό,τι αφορά τώρα την μεταρρύθμιση του κανονισμού 1-2005, επηρεάζεται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τα τέλη που επιβάλλονται για τη μεταφορά εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση των ζώων μέχρι ότου φτάσει το ζώο στην τελικό προορισμό. Και ο κανονισμός αυτός δεν λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή, δεν εφαρμόζεται σωστά και δεν περιλαμβάνει επαρκή προδιαγραφέ για τα οχήματα οι οποίε ούτε επαρκούν ούτε τηρούνται και σε θέματα εκτροφή. Ε, για παράδειγμα. οι παύσεις για την ανάπαυση των ζώων οι οποίες δεν τηρούνται. Κατάρτιζα λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης και ζητώ απαγόρευση όλων των μεταφορών των ζώων που ξεπερνούν τα, τις 8 ώρες και για όταν ο προορισμός είναι το σφαγείο λιγότερο από 4 ώρες ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή και τα σφάγια σε ό,τι αφορά τα ζωντανά ζώα, σε ό,τι αφορά επίσης τους ελέγχους ε, που ζητούμε για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η λογική πίσω από τις προτάσεις μας είναι η εξή. Σε πολλές περιπτώσεις μεταφορών, πολύ απλά δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι κανονισμοί περί μεταφοράς. Και πιστεύω ότι αυτό εξετάζει να το εξετάσουμε. Ε, αυτό αξίζει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Προσβλέπω στη συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Εγώ θα ήθελα να προσθεθούν τρεις τροπολογίες σε τρεις τομείς ουσιαστικά και κάποιες διευκρινήσεις. Οι τομείς αυτοί λοιπόν έχουν να κάνουν με την πυκνότητα των ε, ζώων που μεταφέρονται το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα μικρά και τοπικά σφαγεία και τα κινητά σφαγεία ενδεχομένω. για να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στην επεξεργασία τροφίμων. Και τέλος, να καλέσω για την αναθεώρηση των τελών. Γιατί τα ζώντα ζώα προσελκύουν μάλλον έχουν μια, ένα τέλος 10% ενώ τα σφάγια 40%. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να ισχύει, γιατί αυτό αποτελεί κίνητρο να μεταφέρονται τα ζώα ζωντανά. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την ε, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και οδηγεί σε μεγάλες καταχρήσεις των διατάξεων για την ευημερία των ζώων. Πραγματικά, Αν υπομόνω να ακούσω και την άποψη των άλλων πολιτικών ομάδων. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ. Ο κύριος Βάντεν Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εδώ θα αντικαθιστώ τη συνάδελφο Κλάουντα Μοντερό Αγγελάρη, η οποία εξακολουθεί να είναι σε άδεια μητρότητα. Το είπα και στις 3.30, το ξαναλέω και τώρα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Συμφωνώ με τη βασική προσέγγιση του Κιθ Taylor ότι η ευημερία των ζώων ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τον τομέα των μεταφορών, πόσο μάλλον και για ζώα τα οποία οδεύουν προς το σφαγείο, θα πρέπει να αποτελέσει ένα σημείο εστίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά μεταξύ πρασίνων και ΕΛΚ δεν μπορώ παρά να την εξηγήσω πώς το μεσημέρι. Όποτε υπάρχει πρόβλημα, οι πράσινοι ξαναγράφουν τον κανονισμό για να τον βελτιώσουν θεωρούν. Εμείς, ωστόσο, πιστεύουμε ότι ο κανονισμός του 2005 εξακολουθεί να είναι χρήσιμος και προδιαγράφει με πολύ λεπτόμερη τρόπο το τι θα πρέπει να συμβεί. Πολύ απλά όμως δεν εφαρμόζεται, δεν τηρείται. Τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό. Και η πιο σημαντική συμβολή της Κλάντια Μοντέρο στη συζήτηση αυτή θα είναι να υπάρξει καλύτερη εφαρμόγη του κανονισμού του 2005 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί ως α, θεματοφύλακας. Γιατί και εδώ έχει κάποιες ε, υποσημειώσεις να παρουσιάσει η κυρία Κλάουντια Μοντερό. Μία ερώτηση προς τον κύριο ε, Τέιλορ και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, Πρόεδρε. Ε, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων προσφάτως ανέφερε ότι ο κίνδυνος επιζωοτιών και επιδημιών κατά τη μεταφορά των ζώων δεν είναι τόσο υψηλός όσο θεωρείται. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση της ανάγκης μείωσης του χρόνου μεταφορών. Με άλλα λόγια, εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί καλύτερο ο κανονισμός του 2005 παρά αυτό που λέει ο κύριος Keith Taylor, να καταρτιστούν καινούργιοι κανόνες, γιατί ξέρουμε ότι όταν βάζουμε προδιαγραφές επί προδιαγραφών, ενώ δεν έχουν ουσιαστικά ακόμα εφαρμοστεί και οι προηγούμενε περιγραφέ, είναι σαν να χτίζουμε πάνω στην άμμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Ντεμόντε τώρα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια, κύριε Τέιλορ, για την πρόταση. Είσαστε και πολύ δραστηριο στην ε, διαπαραταξιακή ομάδα για την ε, ευημερία των ζώων, αλλά δεν μου εκπλήσει η εκθεσή σα. Και εγώ είμαι μέλο αυτή τη ομάδα και έχω κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Δεν είμαι σίγουρη ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Πιστεύω ότι η ευημερία των ζώων θα πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητα και όχι τα εμπορικά θέματα. Ε, ειδικά κατά τη μεταφορά ζώων των ζώων, γιατί τα ζώα πέφτουν θύματα καταχρήσεων και οι να εφαρμόζονται σωστά. Αυτό που λείπει πάνω απ' όλα είναι ο αποτελεσματικό έλεγχο. Αυτό καθιστά τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Παρά την, το ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει επικυρώσει τη σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων, τα ίδια κράτη-μέλη δεν σέβονται τους κανόνες. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ενιαίες διαδικασίες, ούτω ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτού του έλεγχου. Είμαι μεταξύ αυτών που υπέγραψαν το αίτημα για να ξεκινήσει μία ε, ερευνητική επιτροπή του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, μια εξεταστική επιτροπή για το θέμα αυτό, δεν είναι δευτερεύον θέμα για μια κοινωνία ή κοινωνίε όπω οι δικέ μα που υποτιθέτουν ότι είναι πολιτισμένε. Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια ήμασταν μάρτυρε ε, πολλών προβλημάτων σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων. Καταρχάς το θέμα που απασχολεί σήμερα είναι το θέμα της μεταφορά ζών των ζώων. Αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Ελπίζω η Κομισιόν, τουλάχιστον για το θέμα της μεταφοράς των ζώων, να δείξει μια, ευελιξη, μια ευαισθησία, κάτι που δεν έχει δείξει τα υπόλοιπα θέματα, θέματα που αφορούν την ε, υγεία και ευμερία των ζώων. Ο κ. Λοτόφσκι έχει τώρα το λόγο. Εγώ ε, εκφράζομαι εξ ονόματος του συναδέλφου μου, τον κ. Λεγκούτκο. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το για τη σωστή εκτίμηση της ε, κατάστασης ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού και την προστασία ζών των ζώων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με τον εισηγητή γιατί η πρόοδος εφαρμογής του κανονισμού του 2005 δεν είναι επαρκής. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ευμερία των ζώων κατά την ε, μεταφορά τους. Κυρίως λόγω του ότι οι κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί ε, δεν είναι αυστηρά τα κράτη-μέλη. Δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Η μεταφορά των ζώων είναι ένα θέμα επίμαχο. Φυσικά είναι αναγκαίο να τα μεταφέρουμε κάποια αυτά τα, κάπως αυτά τα ζώα προς το σφαγείο. Ε, τα ζώα που συμμετέχουν σε αθλητικές ε, δραστηριότητες επίσης και αθλητικούς αγώνες, κάπως πρέπει να τα μεταφέρουμε, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα ζώα να είναι θύματα σκληρότητας. 70 με 80% ε, όλων των μεταφορών των ζώων αφορούν τη μεταφορά ζώων προς τα σφαγεία. Ε, στον κύκλο της εκτροφής ζώων ε, αυτός ο χρόνος μεταφοράς ε, είναι μικρός, αλλά μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τα πράγματα. Αν η, το ταξίδι είναι πολύ μακρύ και κακά οργανωμένο, μπορεί να έχει και επιπτώσεις οικονομικές, αλλά και κακές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι η μεταφορά ε, σφαγμένων ζώων ή κρέατος είναι πολύ πιο αποτελεσματική και είναι και πιο ηθική και σωστή από το να μεταφέρουμε ζώντα ζώα. Η σφαγή των ζώων θα πρέπει να γίνεται σε σφαγεία που βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εκτροφής των ζώων. Η δική μας πολιτική ομάδα θα ήθελε να περιορίσει το χρόνο μεταφοράς των ζώων προς τα σφαγεία σε 8 ώρες, καθώς και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και το χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης. Είτε τα μεταφέρουμε με χερσαίο τρόπο, είτε με θαλάσσιες μεταφορές. Ακόμα και να οργανώσουμε πολύ καλά την ε, μεταφορά το ταξίδι, τα ζώα είναι εγχωμένα και θα πρέπει να μειώσουμε αυτό το στρες. Αυτό εξαρτάται από την ε, εμπειρογνωμοσύνη, τη γνώση του προσωπικού που συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Τα ζώα βγαίνουν από το γνωστό τους περιβάλλον και ήδη αγχώνονται και μόνο, και μόνο να τα φορτώνουμε και να τα ξεφορτώνουμε, τους δημιουργεί τεράστιο άγχος. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να προστατεύει την ευημερία των ζώων κατά τη μεταφορά. Όσο μπορούμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία να έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Keith Τέιλερ για την ε, παρουσίαση της γνωμοδότησης. Το συζήτησαμε και στην ε, προηγούμενη θετία και όντω, ε, όπως είπε ο συνάδελφος Λοτόφσκι, καταρχάς για τα ζώα αυτό που έχει σημασία είναι εφόσον οδεύουν προς το σφαγείο να μην είναι μεγάλη η απόσταση μεταφοράς. Ε, πάντα μιλάμε για την ιστορική αγορά. Αυτό δεν έχει να κάνει όμω μόνο με την ιστορική αγορά. Και εγώ είμαι από την Ήπεθρο και ξέρω ότι υπάρχουν ε, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν λίγα ζώα και βάζουν τις μεταφορές τους μαζί με άλλους, τις οματοποιούν. Και αυτό σημαίνει πολλές ώρες μεταφοράς. Ξέρω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε τρώμε κρέα, σφαγιάζονται λοιπόν τα ζώα και θα πρέπει να σφαγιάζονται και φυσικά αυτές οι μεταφορές είναι κάτι το οποίο δεν μας χαρπεί ιδιαίτερος. Αυτό είναι σαφές. Έχω κι εγώ κάποιες ε, τροπολογίες υπόψη μου για να τις καταθέσω, αλλά Κατά βάση θέλω να πω πώς θα γίνει και αυτή η καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού και τι θα σχολιάσει η, Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Και εγώ θα πάρω το λόγο τώρα από την Επιτροπή μας. Από το 2012. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που γίνονται από τις οργανώσεις υπεράσπισης των ζώων. Και κάθε φορά η ετοιμιγορία είναι καταπέλτης δημιουργούμε τρομακτικές συνθήκες ε, για τη μεταφορά αυτών των ζώων. Η διάρκεια των ταξιδιών, ε, η μέγιστη διάρκεια δεν γίνεται σεβαστή. Παραβιάζουμε 100% την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία έρευνα που κράτησε πέντε χρόνια στα σύνορα με την Τουρκία και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το 2016. Τα αποτελέσματα είναι ανατριχιαστικά. 89% των φορτηγών που μεταφέρουν ε, ζώα από τη Γαλλία παραβίαζαν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2017 και άλλες έρευνες με φορτηγά, με πρόβατα ή αγελάδες, με, με ταβάνια που ήταν πάρα πολύ χαμηλά, που τα κεφάλια των ε, ζώων δεν μπορούσαν να σηκωθούν, δεν είχαν χώρο. Επίσης το σύστημα πότισης και αερισμού δεν λειτουργούσε και οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν κατά πολύ τους 35-40 βαθμούς. Για τις μεταφορές ε, μέσω θάλασσας. Τα σκάφη, ειδικά για τα ζώα, τα οποία είναι ε, εντελώς λάθος σχεδιασμένα, χωρίς κανένα όριο για το ταξίδι. Ούτε ούτε υπάρχει ε, ανάπαυση, ούτε υπάρχει κτηνίατρος ή υπεύθυνο για την προστασία των ζώων ε, του σκάφου. Το σύνολο των ε, ερευνών αυτών έχουν κάποια συμπεράσματα που στηρίζουν την έκθεση ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιστροπής που δημοσιεύτηκε στις 4 Απριλίου που μας πέρασε για μη συμμόρφωση ε, πάνω από το 5% των περιπτώσεων και φοβερά κενά σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των ζώων. Ε, ειδικά κατά τη μεταφορά ζώων προς το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι σκάνδαλο. Και το λέω εδώ επίσημα στην Επιτροπή μας. Εφεξής, θα πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες είναι απάνθρωπες, σκληρές που υφίστανται τα ζώα. Τα ζώα δεν θα πρέπει να υποφέρουν. Δεν θα πρέπει να περνάνε όλα αυτά που τα αναγκάζουν να περάσουν. Ε, θα πρέπει να βάλουμε τέλος αυτήν την ιστορία. Γιατί υποφέρουν περιτά. Γιατί δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Είναι και η ώρα να βελτιώσουμε την ζωή των ζώων, την ευημερία τους, αλλά κυρίως να θέσουμε και εμείς κάποια ερωτήματα στον εαυτό μας. Πώς γίνεται και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την καταστροφική κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σας, ε, κυρία Ντεμόντε, ότι η κατάσταση κατά τις μεταφορές ε, θα έπρεπε να μας οδηγήσει στη σύσταση μιας πραγματικής κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής. Τώρα όμως έχουμε αυτή την έκθεση. Θα την ε, ολοκληρώσουμε, θα είναι φιλόδοξη, ούτως ώστε να σημαδέψει τους πάντες. Θέλω να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you very, very much, uh, Madam. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Τέιλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι δεν πρέπει να υποφέρουν τα ζώα κατά τη μεταφορά τους. Ωστόσο, δεν συμφωνεί με αυτό που περιγράψατε, ότι δηλαδή οι μεταφορέ των ζώων στην Ευρώπη είναι καταστροφή, μια καταστροφική κατάσταση, μια δραματική κατάσταση. Έχουμε νομοθεσία και έχουμε και στοιχεία. Εάν δούμε τα στοιχεία αυτά, μας δείχνουν ότι έχουμε εκατομμύρια μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότερες από αυτές γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία. Πρέπει να ενισχύσουμε την ε, υφιστάμενη νομοθεσία γιατί πράγματι μπορεί να βελτιωθεί. τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα αυτών. Προσπαθούμε ε, και εργαζόμαστε και στον τομέα των οδικών μεταφορών και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ε, να έχουμε ομάδες στα κράτη-μέλη με, τις οποίες συνερ... Ε, με τις οποίες παρακολουθούμε αυτές τις μεταφορές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοσιοποιήσουμε εκθέσεις και για την κατάσταση μέσω των οδικών μεταφορών και για την κατάσταση όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Επίση, μια και αναφερθήκατε σε κάποια στοιχεία, θα ήθελα να μα τα κοινοποιήσετε, γιατί είναι λανθασμένο κατά την άποψή μα κάποιο να ξεχωρίζει τι ε, αρνητικέ περιπτώσει, τα άσχημα παραδείγματα και να τα βλέπει εκτό του πλαισίου του. Εγώ πιστεύω ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν χρειάζεται να ε, υποφέρουν ανεφλόγου στα τα ζώα και η υφιστάμενη νομοθεσία μας το εξασφαλίζει. Αυτό πρέπει βέβαια να βελτιωθεί η Πρόεδρος. Κύριε Τέιλορ, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ μαζί σας ότι το 97% των μεταφορών των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρεί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Αυτό δεν είπατε, αυτό είπατε. Ε, έτσι το κατάλαβα εγώ, έτσι φαντάζομαι το κατάλαβαν και οι συνάδελφοι. Πάντως αυτό δεν ισχύει, δεν είναι αλήθεια. Όπως ήδη ανέφερε η Πρόεδρος, έχουμε καταγράψει ότι 3 εκατομμύρια ζώα εξήχθησαν, εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τρίτες χώρες με ε, ε, κατά συνθήκες μεταφοράς οι οποίες είναι απάνθρωπες και ε, απαράδεκτες και ακόμα χειρότερες, χειρότερη μεταχείριση όταν φτάσουν πια στον προορισμό τους. Ο κύριος Βαντερκάμπ μας λέει ότι ο κανονισμός είναι απαρκής. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι δεν εφαρμόζεται. Ναι, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα πρότυπα που υιοθετούμε. Δεν λέω κάτι καινούριο. Αυτό που λέω ουσιαστικά είναι ότι θα πρέπει να δούμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακολουθήσουμε το σκεπτικό της όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων. Χαίρομαι τουλάχιστον που από πολλού συναδέλφου υπάρχει η αναγνώριση του ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Και είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε και μια πολύ καλή συνεργασία με τα μέλη από τι επιτροπέ ΕΝΒΙ και ΆΓΡΙ έτσι ώστε να αναλάβουμε δράση για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Προθεσμία ε, κατάθεση των τροπολογιών 27 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Εάν δεν υπάρχει κάποιο θέμα υπό τα διάφορα, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018. Εν τω μεταξύ, καλό απόγευμα. Allez